Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Καθίστε παρακαλώ. Είναι παρόντες και οι συγητέ μας. Αρχίζουμε με λίγα λεπτά καθυστέρηση. Είναι πολύ φορτωμένο όμως το πρόγραμμά μας σήμερα και θα σας παρακαλούσα να καθίσετε διότι δεν έχουμε και υπερβολικό χρόνο και καλό θα ήταν να αρχίσουμε λοιπόν. Και εξ ονόματος του συναδέλφου κυρίου Ντανζάν ε, που είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής Αμήνης. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή τη δεύτερη διακοινοβουλευτική συνέλευση της χρονιάς. Θα θυμάστε η προηγούμενη ε, συνεδρίαση ε, αφορούσε στις 2 Ιουνίου ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σήμερα θα θέλαμε να αφιερώσουμε τη συνάντησή μας σε ένα θέμα εξαιρετικού ενδιαφέροντος για όλους μας. Είναι προκλήσεις, αλλά όχι μόνο προκλήσεις, αλλά και οι ευκαιρίες, θα έλεγα, που προσφέρει στην ΚΕΠΑ η συνθήκη της Αβώνας στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία και στην ε, ΕΠΑ που είναι Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλεία και Αμυνα. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τον κύριο Σαστέλ ε, που είναι εδώ υπό την ιδιότητα του προσώπου της ε, Βαρόνης Άστον που είχε σήμερα ανηλυμένε υποχρεώσεις γιατί συναντά τους Αμερικανούς ομολόγου τη και θα ακούσουμε και τον Υπουργό Ντεκρέμ, Υπουργό Αμήνη του Βελγίου στη συνέχεια. Ε, τελικά όμως ε, δεν θα έρθει και τον εκπροσωπεί ο κύριο Αστέρ. Λοιπόν, εκπροσωπούνται όλα τα κοινοβούλια εκτός από τη Βουλή των Κατοχωρών και τη Βουλή της Τσεχική Δημοκρατίας. Στόχος μας είναι να δώσουμε μια ισχυρή ε, κοινοβουλευτική διάσταση στην πολιτική αυτή. Η σημερινή συνεδρίαση θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε όλοι μαζί ε, για τις αλλαγές λοιπόν που ε, επιφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στα πλαίσια διαφόρων άλλων δράσεων και σενάριων. Γι' αυτό σας απευθύνθηκε η πρόσκληση αυτή καθώς επίσης και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν, που είναι κρίσιμη η περιοχή, και θα μιλήσουμε και για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Και το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει παρουσία εκπροσώπου του. Ελπίζω ε, στο τέλος της συνεδρίασης να έχουμε ξεκαθαρίσει λίγο στο μυαλό μας τα πράγματα και να έχουμε καταλάβει ποιες είναι οι αμοιβέ μας ευθύνες και αρμοδιότητες και εσάς των Εθνικών Βουλευτών και εμάς των Ευρωβουλευτών. Λοιπόν, η διάσκεψη των Προέδρων των ε, Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισε μια τέτοια προσπάθεια για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ελπίζω να είναι και χρήσιμη και επικοδομητική η σημερινή συνεδρίαση. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο και συμπρόεδρο κύριο Ντόρζαν. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω εξ ονόματος Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αυτή τη συνεδρίαση, τη συνάντηση, όπως θύμισε ο πρόεδρος Αλμπερτίνη, ξεκινάμε μια πολύ χρήσιμη και σημαντική συζήτηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια για την εφαρμογή των νέων διατάξεων της Συνθήκης Λισαβόνας στον τομέα της, πολι... της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι αυτή η συνθήκη επιτρέπει ένα άλμα προς τα μπρος περνάμε από την ΚΕΠΑ στην ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας που θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικές ρήτρε οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στην κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πραγματοποιήσει ένα πραγματικά ποιοτικό άλμα. Αυτή η συνθήκη, θα ήθελα να σας θυμίσω, προβλέπει τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, είπα, του, εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική της ε, κοινότητας με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης μια ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας και μια ρήτρα αλληλεγγύης δύο στοιχεία πολύ καινοτόμα και σημαντικά την επέκταση των αποστολών στην, ε, που αναλαμβάνει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, μόνιμες επιτροπές και δομές για τις χώρες που έχουν πιο μεγάλη στρατιωτική ικανότητα και αναλαμβάνουν σε αυτό το τομέα πιο δεσμευτικές υποχρεώσεις και ένα ταμείο χρηματοδότησης για τις παρασκευαστικές ε, για τη χρηματοδότηση των προπαρασκευή της προπαρασκευής των διαφόρων δράσεων. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε μαζί στα πλαίσια της ε, κοινοβουλευτική κοινοβουλευτικής παρακολούθησης των εξελίξεων και είμαι βέβαιος ότι οι σημερινές μας συζητήσεις θα αποδειχθούν ιδιαίτερα καρποφόρες. Σεστέλ. Η συνθήκη της Λισαβόνας εξασφαλίζει τη συνεργασία στην Ευρώπη σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Αυτό συμβαίνει την εποχή που η ευρωπαϊκή κοινότητα καλείται να δώσει εγγυήσει για την ασφάλεια και την άμυνα. Ταυτόχρονα η ασφάλεια, η άμυνα και η σταθερότητα απαιτούν την ε, εμπλοκή, τη συμμετοχή πολιτικών δομών, ενώ η στρατιωτική ε, ικανότητα προσανατολίζεται ε, στην διεξαγωγή πολιτικών αλλά και στρατιωτικών αποστολών. Η οικονομική κρίση σημαίνει επίσης ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εξορθολογήσουν τις δαπάνες τους και αυτό γίνεται με σημαντικές περικοπές στο προϋπολογισμό για την άμυνα σε πολλές περιπτώσεις. Η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης επιδιώκει ε, ε, να βρει συνέργειες, κάτι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαστέλ που ήρθε να μας συναντήσει σήμερα το πρωί και θα του δώσω το λόγο για να μας μιλήσει για τις δυνατότητες που μας προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας να αναδιατυπώσουμε μια κοινή εξωτερική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας η οποία να είναι συνεπής με τους στόχους της συνθήκης. Όταν οι συνάδελφοι θα παίρνουν το λόγο, τους παρακαλώ να είναι σύντομοι και θα παρακαλέσω τον κύριο Σαστέλ να δώσει το παράδειγμα χρησιμοποιώντας για την ομιλία του όχι παραπάνω από 15 λεπτά. Οι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο καλούνται να συμπληρώσουν ένα μικρό δελτίο που έχουν στο μπροστά του για να τα συγκεντρώσουμε και να οργανώσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Αστέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλη των Κοινοβουλίων των 27 κρατών μελών, αγαπητοί συνάδελφοι, για μένα είναι πραγματική χαρά που απευθύνομαι ε, σήμερα εξ ονόματο τη ΣΥΠΑ της εκπροσώπου τη κυρία Κάθριν Άστον σε αυτή την πρώτη διακοινοβουλευτική συνάντηση για την κοινή πολιτική Άμυνα και ασφάλεια ασφάλειας. Ο Βέλγος συνάδελφός μου για την άμυνα, ο υπουργό Πίτερ Ντεκρέν, θα ήθελε ασφαλώς να είναι, θα ήταν ασφαλώς ένας πιο κατάλληλος ομιλητή για να μιλήσει εξ ονόματος της ΥΠΑ εκπροσώπου για αυτό το θέμα. Αλλά δυστυχώς εμποδίστηκε, δεν, είχε, δεν μπόρεσε να έρθει και γι' αυτό μου ζήτησαν τον αντικαταστήσω. Αυτή η διάσκεψη λαμβάνει χώρα σε μια σημαντική στιγμή. Την 1η Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί, περάσει ένα χρόνο από την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ορισμένε από τι νέε διατάξει που προβλέπει η συνθήκη εφαρμόζονται ήδη, παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά το ρόλο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του ΙΠΑ του εκπροσώπου. Άλλε διατάξει πρέπει να εξεταστούν πιο προσεκτικά και να αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνία για να εφαρμοστούν. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα καταστεί λειτουργική σε λίγου μήνε, θα συγκεντρώσει στην ίδια δομή τα διάφορα μέσα και τι διάφορε υπηρεσίε εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτέ που συνδέονται με την πολιτική, πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Μιλάμε για ουσιαστική πρόοδο, για ουσιαστικό βήμα προ τα μπρο και αυτή η υπηρεσία είμαι βέβαιο ότι θα δώσει νέα όθηση στη δράση μα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση είναι ένα από τα νέα μέσα που προβλέπει η συνθήκη τη Λισαβόνα για την ενίσχυση της συνοχής και της αποφασιστικότητας των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εξωτερικό επίπεδο και θα συμβάλλει στην ανάληψη της ε, κοινότητα της Ένωσης όλο και πιο σημαντικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Αντιμετωπίζουμε βεβαίως και τις φοβερές συνέπειες της οικονομικής κρίσης και ως υπεύθυνοι για την πολιτική καλούμαστε να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις για να αποφασίσουμε πού θα περικοπούν οι δαπάνε και οι δαπάνε για την άμυνα δεν είναι βεβαιω δυνατόν να μην περιληφθούν σε αυτά τα μέτρα. Σε όλε τι κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κοινοβούλια και οι αρμόδιες επιτροπέ για την εξωτερική πολιτική και τα θέματα τη άμυνας και τη ασφάλεια συζητούν αυτό το θέμα. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την διακοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα τη κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια, επιτρέποντα τα κοινοβούλια να ανταλλάσσουν απόψει και εμπειρίες συνεργασίες μεταξύ τους. Η βασική πρόκληση για τους Υπουργούς Άμυνας είναι να δουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση στην Ευρώπη εφαρμόζοντα μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να βρούμε τα μέσα, να δαπανάμε πιο αποτελεσματικά τα χρήματά μας, να αξιοποιούμε πιο σωστά τους πόρους που διαθέτουμε για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, θα χρειαστεί να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας. Η βελτίωση των ικανοτήτων θα οπωσδήποτε θα ε, φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς στους οποίους διαθέτουν πόρους οι διάφορες χώρες σε εθνικό ή ε, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο. Πρέπει να συσπυρώσουμε τις προσπάθειες και τις δυνάμεις μας ως Ευρωπαίοι και να αξιοποιήσουμε τα ισχυρά μα σημεία. Στη Γάνδη έγινε μια συζήτηση πριν εβδομάδα μεταξύ Υπουργών Άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που, που συνεδρίασαν σε άτυπο συμβούλιο. Επί τη ουσία επετεύχθη σύμπτωση απόψεων κρίναμε ότι πρέπει να επιδείξουμε ουσιαστική αποφασιστικότητα, να αντλήσουμε διδάγματα από τις, από τις εμπειρίες μας και να ε, ενώσουμε τις προσπάθειές μας. Αν μπορέσουμε να δώσουμε σωστές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι καλύτερα στη θέση να παίξει το ρόλο της στον τομέα της ασφάλειας, να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις που αυξάνονται και να απαντήσει στις προσδοκίες των πολιτών οι αποφάσει για τον τρόπο να περιοριστούν οι δαπάνε για την άμυνα σε εθνικό επίπεδο λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τι ε, οικονομικέ ανάγκε. Στη Γάνδη, σε αυτό το άτυπο συμβούλιο ωστόσο, οι υπουργοί συζήτησαν επίση το γεγονό ότι αυτή η απόφαση θα πρέπει να καθοδηγείται από μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση και σύλληψη του κοινού στόχου που πρέπει να επιτευχθεί και των μέσων για την επίτευξή του. Μπορεί να χρειαστεί να περιορίσουμε το μέγεθο των ε, ενόπλων δυνάμεών μα, Αν λάβουμε από, από κοινού τις σωστέ αποφάσεις θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Όταν μιλάμε για τα μέσα να επιτύχουμε αυτό το στόχο, τα μέσα για να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την ικανότητα δράσης της Ευρώπης, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για ευρύτερη συνεργασία μεταξύ μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι η συνεργασία στον τομέα της άμυνας είναι ένας δύσκολος θέμα, διότι αγγίζει σημαντικά στοιχεία ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Ωστόσο μπορεί να ενέχει και σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρέπει να συνεργαστούμε για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη δυναμικότητα την οποία χρειαζόμαστε και να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες για οικονομίες κλίμακας. Μπορούμε επίση να περιορίσουμε το κόστος ε, ε, εφόσον μοιραστούμε και χρησιμοποιούμε από κοινού τις υπάρχουσες ικανότητες, δυναμικότητες σε ευρωπαϊκό ενωσιακό επίπεδο ή στο, σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο. Όλοι γνωρίζουμε τι χρειαζόμαστε. Πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Ένα σημαντικό παράδειγμα μας παρέχεται από την ε, υπηρεσία ε, πολιτικής αεροπορίας στο Eindhoven που συντονίζει τις ε, αεροπορικές μεταφορές της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας. Μπορούν να συμμετάσχουν και άλλες χώρες. Αυτή η δομή θα αξιοποιήσει τις ικανότητες για τις εμπορευματικές αεροπορικές μεταφορές, επιτρέποντάς μας να, συνδυάσουμε, να συνδυάσουμε τις δράσεις μας σε θέατρα πολέμου όπως είναι το Αφγανιστάν. Έτσι θα ξεκινήσει μια συνεργασία και καλύτερη αναρμόνιση στον τομέα των στρατηγικών αεροπορικών μεταφορών. Η συνθήκη της Αβώνας προβλέπει όχι μόνο τα κράτη-μέλη θα βελτιώσουν τη δυναμικότητά τους για να υποστηρίξουν την ΚΕΠΑ αλλά και, την πολιτική άμυνας και ασφάλειας αλλά και μόνιμες δομές που θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη που επιθυμούν να επεκτείνουν και να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας να οργανωθούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συζητήσει που είχαν σκοπό να καταλήξουν σε μια ερμηνεία κοινή των διατάξεων της συνθήκης συνεχίζονται. Αυτό αποτελεί ένα πρώτο στάδιο, μια πρώτη φάση και γι' αυτό το λόγο ένα σεμινάριο στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών έγινε, έλαβε χώρα τον περασμένο Ιούλιο το άνοιγμα, η εξωστρέφεια είναι η λέξη κλειδί. Πρέπει να εξασφαλίσουμε απόλυτη διαφάνεια και μεγάλο βαθμό ευελιξίας αλλά θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για να καθορίσουμε ποιες δομές που δεν υπάρχουν ήδη στο πλαίσιο της Ένωσης θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για να ενισχύσουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις ακόμα και στον Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας αυτή η ανα, των ικανοτήτων είναι σημαντική, διότι χωρίς ικανότητες δεν μπορεί να υπάρξει εξωτερική, ε, ε, ευρωπαϊκή πολιτική, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές και τις μελλοντικές κρίσεις. Η ικανότητα δράσης της Ένωσης θα ενισχύσει τον πολυμερισμό και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και στην προώθηση της ειρήνης και του κράτους δικαίου οι προκλήσει στι οποίε οποίες καλούμαστε να απαντήσουμε σήμερα, παραδείγματο χάρη στο Αφγανιστάν και στη Σομαλία, είναι τεράστια. Τα σενάρια κρίσης είναι σύνθετα. Αδύναμα, ε, αδύναμες κυβερνήσεις, αδύναμα κράτη που δεν μπορούν να ελέγχουν την επικράτειά τους, έλλειψη δημοκρατικών δομών, ε, διαφθορά, ατιμορρησία γενικευμένη, ομάδες που αγωνίζονται για την εξουσία και τους πόρους, δυστυχία των πολιτών που είναι τα κύρια θύματα. Αν πρέπει να, για να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα πρέπει να αποφύγουμε οι κίνδυνοι σε θέματα ασφάλειας που εκπροσωπούν αυτές οι περιοχές να μην θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ευρώπης. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν ε, απλές απαντήσεις που θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε σε αυτές τις κρίσεις και να εγγυηθούμε τη σταθερότητα και ότι πρέπει να εξετάσουμε όλο το φάσμα των μέσων που διαθέτουμε. Διπλωματία, ανάπτυξη, οικονομία, ε, ανάπτυξη πολιτικών και στατιωτικών μέσων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα διαθέτει όλα αυτά τα μέσα και η συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε τη δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα χρησιμοποιεί όλα αυτά τα μέσα με συντονισμένο τρόπο. Όταν ο σεισμός της ΑΕΤΙΣ επήλθε και μας το θύμισε, δεν αρκεί να διαθέτουμε μέσα και εργαλεία για να αντιδράσουμε με αποτελεσματικό και κατάλληλο τρόπο. Χρειάζεται επίσης συντονισμός βέλτιστο δυνατό συντονισμό. Σε λιγότερο από 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε πάνω από 20 αποστολέ διαχείριση κρίση σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Η δράση των αποστολών ενισχύεται συχνά και στηρίζεται από άλλα μέτρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διπλωματικά μέσα όπω οι ειδικοί εκπρόσωποι τη Ένωση, η χρηματοδότηση συμπληρωματικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δουλεύουμε σε στενή συνεργασία με του εταίρου μα και βεβαίω με τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και το ΝΑΤΟ και πολλούς άλλους οργανισμούς επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα παραδείγματα. Στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, στο Κόσοβο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οργάνωσε διπλωματικές οικονομικές αποστολές υπέρ της σταθερότητας και για μια ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών αυτών. Οι δικοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβαν να συνοδεύσουν εξ ονόματος τη διεθνούς κοινότητας τις μεταρρυθμίσεις που είχαν ξεκινήσει σε πολιτικό επίπεδο. Ε, επιχειρήσεις ε, διαχείρισης κρίσεως συνέβαιναν στην δημιουργία ενό ασφαλού περιβάλλοντος επιτρέποντα στις τοπικές αρχές να εγγυώνται το κράτος δικαίου άλλες δράσεις για την καταπολέμηση της πειρατεία, τα νυχτά τη Σομαλίας βρίσκεται στο επίκεντρο της ε, βούλησης της ε, Ένωσης και της, Ευρωπαϊ... και διεθνούς κοινότητας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της πειρατείας με αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με τις θαλάσσιες μεταφορές, εφαρμόστηκαν ευρύτερα προληπτικά μέτρα για το συντονισμό με τις άλλες ναυτικές δυνάμεις που είναι ανεπτυγμένες στην περιοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε συμφωνή με τις γειτονικές χώρες για τη μεταφορά των συλληφθέντων πειρατών. Η βοήθεια που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις χώρες είχε σκοπό να ενισχύσει τη δυνατότητά τους να συλλαμβάνουν και να φυλακίζουν τους υπόπτους και να ε, εξασφαλίσουν για χρηστή διακυβέρνηση σε αυτό το τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει συζητήσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για την ανέβρεση μιας μόνιμης λύσης σε ό,τι αφορά την ε, παρακολούθηση και σύλληψη των υπόπτων για πειρατεία. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σκοπεύει να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της ε, πειρατείας η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύοντας τις δυνατότητες των χωρών της περιοχής. Έχουμε προγράμματα κατάρτισης στην Ουγγάντα για την προετοιμασία των δυνάμεων της Σομαλίας και τη συμμετοχή τους σε, παγκόσ... σε διεθνείς δράσεις ώστε το κράτος της Σομαλίας που είναι αποδυναμωμένο να μπορεί τουλάχιστον να ασκεί την εξουσία στην επικράτειά του. Υπάρχουν προγράμματα για την παροχή βοήθειας τη ευρωπαϊκή Ένωση, για την ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή. Ο απολογισμός των δράσεών μας είναι εντυπωσιακό. Βεβαίως πάντοτε δεν καταφέραμε να λύνουμε τα προβλήματα αυτά αλλά η δράση μας είχε απτά αποτελέσματα, ενώ η ικανότητα και οι δυνατότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης σαφώς αποδείχθηκαν. Η συνθήκη της Λισαβόνας με τη δημιουργία της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θα είναι το εργαλείο που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες αυτές με βάση την αποκτηθή σαπήρα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεν θα αλλάξει τους μηχανισμούς και τα μέσα στον διπλωματικό ε, και οικονομικό κόσμο και στη διαχείριση κρίσεων, αλλά θα υποστηρίξει την εφαρμογή συνεκτικών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προλαμβάνουμε κρίσεις και να χρησιμοποιούνται τα μέσα κατά συντονισμένο τρόπο και να ενισχύονται. Οι αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασχοληθούν με θέματα εξωτερικής δράσης in situ και θα προσπαθήσουν να ε, σταθούν στο ύψος των αποστολών μας. Η συνθήκη της Λισαβόνας και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επιτρέπει την ενίσχυση της ΕΠΑ και επίσης την ενίσχυση και τον συντονισμό, τον εσωτερικό συντονισμό του στρατιωτικού και πολιτικού σκέλους συνεργασίας στον τομέα της άμυνας. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες καταστάσεις όπου η διαχείριση κρίσεων σημαίνει ότι πρέπει να γίνει χρήση και του στρατιωτικού και του πολιτικού σκέλους, βλέπουμε ότι και το Αφγανιστάν και η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό καταδεικνύουν σαφώς αυτό το παράδειγμα. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε μια κυβέρνηση στη σύσταση της ε, μιας αστυνομίας, ενόπλων δυνάμεων, καθώς και κοινωνικών δομών και την βοηθήσαμε στην αναπτυξιακή της πολιτική. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ε, δύσκολες και περίπλοκες καταστάσεις θα πρέπει να υπάρχει σωστή προσέγγιση πρωτίστως και θα πρέπει να διαθέτουμε στρατιωτικές και πολιτικές δυνάμεις. Πιστεύω ότι οι πολίτες μπορούν να ευεργετηθούν από τις στρατιωτικές δομές και το στρατιωτικό σκέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υποδομές του πολιτικού. Ήδη έχουμε προοδεύσει σε αυτό το τομέα. Προωθούμε τις συνέργειες μεταξύ της ανάπτυξης στρατιωτικών και πολιτικών ικανοτήτων για να υπάρχει διπλή χρήση και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις στρατιωτικές και πολιτικές απόστολες, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της κάθε μίας. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να εξασφαλίσουν τη σωστή κατάρτιση και εκπαίδευση, έτσι ώστε το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό να μπορέσει να ανταποκριθεί στα υψηλά του καθήκοντα. Τέλος, η συνθήκη της Λισαβόνα προβλέπει ρητά να υπάρχει συντονισμός των στρατιωτικών και πολιτικών δράσεων μέσα στα πλαίσια της ΕΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα αφορά τη διαχείριση κρίσεων, με συγχωρείτε, με το πολιτικό, με συνεργασία πολιτικού και στρατιωτικού σκέλους στα πλαίσια της ανάπτυξης των στρατιωτικών και πολιτικών ικανοτήτων. Συνάδελφοι, μίλησα για την ε, συνετή χρήση των στρατιωτικών ικανοτήτων σε συντονισμό με άλλα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα τώρα να σταθώ στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις. Η συνεργασία με τους εταίρους ήταν ένα από τα θεμέλια της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί έναν από τους πυλώνες των πολύπλευρων, των πολυμερών σχέσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι οι εταιρικές αυτές σχέσεις αποτελούν ε, θεμέλιο λίθο της δράσης μας μέσα στον χαρακτήρα της συμπληρωματικότητας όπου θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα από κοινού και θα καταβάλουμε κοινέ προσπάθειες αντιμετώπισης κρίσεων. Το Σεπτέμβριο, μέσα στα πλαίσια του, της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τη συνθήκη της Λισαβόνας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε συντονισμένα τις κοινέ προκλήσεις και να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του διεθνούς προσκυνίου. Άρα η εταιρικότητα αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής και κοινή δράσης. Η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη είναι ακρογωνιας λίθος της συνεργασίας μας και ξέρουμε ότι πέρα από τις ε, επίσημες και πανηγυρικές δηλώσεις θα υπάρχει στενή συνεργασία επιτόπου. Μέσα στα πλαίσια της ε, μέσα στα πλαίσια της αντιμετώπισης κρίσεων υπάρχει μία δύναμη κρούσης, θα υπάρχουν δυνάμεις κρούσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με βάση την ULEX στο Κωσυφοπέδιο και την αντίστοιχη δύναμη κρούσης στο Τσάντ. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή τη συνεργασία. Και το προσωπικό και των δύο οργανώσεων θα ανταποκριθεί σε αυτό το έργο με βάση την κοινή δήλωση του 2003 για την κοινή διαχείριση κρίσεων και τη δήλωση του 2007 για τη συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαχείριση κρίσεων. Θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία όπως, κατέδειξαν η, όπως κατέδειξε η μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο οργανισμών, διότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν εντελώς διαφορετικό τρόπο διαχείρισης. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία μέσα στα πλαίσια και της δράσης των Ηνωμένων Εθνών. Μέσα στα πλαίσια της ΕΠΑ, ένας άλλος ε, ακρογωνιαίος λίθος είναι και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Οι δύο οργανώσεις εργάζονται από κοινού στη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κωσυφχοπέδιο και Αφγανιστάν, καθώς και στις ακτές της Σομαλίας. Σημεριζόμαστε τις ίδιες αξίες και έχουμε κοινού στόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να συντονιστούν όπως δεν προβλεπόταν αρχικά από το αρχικό από την αρχική, πρωταρχική λειτουργία των δύο οργανώσεων. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την εταιρικότητα. Το Σεπτέμβριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την ύπατη εκπρόσωπο να αναφέρει πώς μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ με βάση συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουν διαβιβαστεί στο ΝΑΤΟ στην αρχή του έτους. Προβλέπουμε διαβουλεύσεις και επαφές για θέματα ανάπτυξης πολιτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων έτσι ώστε να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία. Αυτή η διτή προσέγγιση θα συνεχιστεί κατά τους επόμενους μήνες και όλοι οι εταίροι στα δύο αυτά όργανα έδειξαν ενότητα στην αντιμετώπιση των θεμάτων που μας απασχολούν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Το ΝΑΤΟ θα προβάλλει το στρατηγικό του ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προωθήσει τη συνεργασία και με τον πρόεδρο Ομπάμα. Επίσης θα πρέπει να δούμε τις αναδυόμενες δυνάμεις μέσα στα πλαίσια των διεθνών οργανώσεων για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε θέματα κρίσης. Αυτοί οι φορείς αναγνωρίζουν την σημασία του στρατηγικού ρόλου του αναπτυσσόμενου στρατηγικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διαπιστώνουμε στα πλαίσια καταπολέμησης της πειρατείας, όπου αρχίσαμε μία συνεργασία με χώρες που δεν ήταν εταίροι στη διαχείριση κρίσεων, όπως Ινδία, Κίνα και Ιαπωνία αντιμετωπίζουμε την πειρατεία και με τις χώρες ασεάν όπως καταδεικνύει η συνεργασία ευρώπης ασίας η λαϊκή δημοκρατία του κονγκό η κίνα και η νότιος αφρική αποτελούν ένα άλλο απτό παράδειγμα. η συνεργασία με τη ΣΥΠΑ αποτελεί μια πραγματικότητα και η στρατιωτική συνεργασία στο τσάντ κατέδειξε την ύψιστη τη σημασία συνεργασίας με τη ρωσία. οι προοπτικές για την ΕΠΑ ενισχύονται και πολλαπλασιάζονται, όπως ε, δείχνουν και οι χρηματοοικονομικοί πόροι. Θα πρέπει να προβάλλουμε μια πολιτική συνεργασία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προβλέπει ενίσχυση του ενδοκινοβουλευτικού διαλόγου, όπως ε, προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση δεν θα συνεχίσει να υφίσταται. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας διακοινοβουλευτικός διάλογος για να δώσει συνέχεια σε αυτή τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προβάλλουμε μια, έναν κοινό πολιτισμό άμυνας και ασφάλειας. Άρα τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό θα ορίσουν αυτή τη συνεργασία όπως προβλέπει το πρωτόκολλο υπαριθμών 1 της συνθήκης και όπως δήλωσε και η διάσκεψη των προέδρων των ΙΠΕΞ που συνήλθε στη Μαδρίτη την Άνοιξη. Η ύπατη εκπρόσωπος, η κυρία Άστον, θα διευκολύνει τον διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια τα οποία θα μπορούν να, συμμετέχουν, να συμμετάσχουν στις 18 Οκτωβρίου στην ΑΦΕΤ και στην Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης στις 27 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριοι εκπρόσωποι των 27 κρατών μελών, πριν ολοκληρώσω θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να τιμήσω τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν σε αυτή τη συνεργασία ανά τον κόσμο. Ο επαγγελματισμός τους στα πλαίσια των διαφόρων αποστολών δείχνει ότι μπορούμε να προβάλλουμε μία αγαστή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Εθνών και Εθνικής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ε, διεξοδική η παρέμβασή σας. Ζήτησαν το λόγο πολλοί συνάδελφοι και θα τους δώσω το λόγο. Ο κύριος Λεονκέρες που εκπροσωπεί τη γερουσία της ε, Πολωνίας. Ο κύριος Κέρες έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Σαστέλ. Πολύ χρήσιμη η παρουσίασή του και μας εφιστά την προσοχή σε τρεις βασικές παραδοχές. Στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε μια συναντήληψη όλες οι χώρες για τη συνεργασία μας, για την αμοιβαία υποστήριξη και ε, συνδρομή και ε, για ε, τη ρήτρα αλληλεγγύης και υποστήριξης. Βλέπουμε ότι έχουμε νέες δυνατότητες τώρα και ε, μια ομάδα κρατομελών μπορεί να συμμετέχει σε μια κοινή αποστολή. Θα ήθελα λοιπόν, όχι μόνο εξ ονόματός μου, αλλά και εξ ονόματος της γερουσίας της πολωνικής δημοκρατίας, θα ήθελα να ε, σας ευστήσω την προσοχή ε, στο εξής σημαντικό, που έχει σχέση με ένα κοινό ορισμό. Θα πρέπει από κοινού να ορίσουμε τη διαρθρωμένη συνεργασία. Η διαρθρωτική συνεργασία. Ο κύριος Αστέλ μόλις είπε ότι δεν ε, μας φτάνουν τα μέσα και τα εργαλεία ε, που να μας δίνουν τη δυνατότητα αυτή. Θα πρέπει να ξέρουμε και πώς να τα συντονίζουμε. Έτσι λοιπόν έχω την αίσθηση ότι για να ε, είναι δεδομένος αυτός ο συντονισμός των διαφόρων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, θα πρέπει από την αρχή να ορίσουμε τι θέλουμε, ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτής της συνεργασίας, τι κρύβεται πίσω από τα εργαλεία αυτά. Ποια είναι η κεντρική ιδέα. Δηλαδή, από τον ορισμό θα πρέπει να ξεκινήσουμε, να συμφωνήσουμε ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι μαζί το ίδιο όταν λέμε ε, διαρθρωτική συνεργασία. Μετά, η ρήτρα αμοιβαία συνδρομή. Για μένα είναι θεμελιώδου σημασία. Γιατί όλο και περισσότερο εξαρτώμεθα ε, από ε, διάφορους παράγοντες. Θα πρέπει, επαναλαμβάνω, όλοι μαζί να έχουμε την ίδια αντίληψη για το τι σημαίνει η ρήτρα αμοιβαία συνδρομής, τι σημαίνει η διαρθρωμένη συνεργασία, πώς θα συμμετέχουμε σε κάποιες δράσεις. Όταν ε, ε, συμμεριζόμαστε και, και μοιραζόμαστε και κοινέ αποστολές και στρατιωτικές. Άρα θα πρέπει να μοιράζεται και το κόστος και η συμμετοχή του καθενός. Και θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 42 και στο άρθρο 44 της συνθήκης που ορίζει ότι μια ομάδα κρατών μελών μπορούν να ε, αναλάβουν μια συγκεκριμένη αποστολή που θα τους έχει ανατεθεί. Έτσι μια ομάδα κρατών μελών αναλαμβάνουν ευθύνη για μια συγκεκριμένη δράση. Είναι το άρθρο 42 και το άρθρο 44 που βρίσκει ε, άμεση εφαρμογή από τα κράτη-μέλη και είναι ιδιαίτερη αυτή η διάσταση και η πρόκληση. Επαναλαμβάνω, ε, δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου λέγοντας αυτά μόνο, αλλά και το σύνολο της γερουσίας ε, της Πολωνίας. Να δούμε πώς θα τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, καλές οι διατάξεις, αλλά να έχουμε ενιαία αντίληψη για το τι εστί αυτό και τι ορίζει η συνθήκη της Λισαβόνας. Τα άρθρα αυτά που ανέφερα δεν θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν συνεννοηθούμε και συμφωνήσουμε τι εννοούν. Τι σημαίνει ότι αναθέτουμε μία αποστολή σε μία ομάδα κρατών μελών. Τελειώνοντας, θα ήθελα επίσης να πω ότι η Πολωνία υποστηρίζει στεναρά και ειλικρινά την προσέγγιση που ε, μόλις ε, περιέγραψε ο κύριος Σαστέρ. Θέτουμε το κέντρο βάρους στη βούληση πραγματικά των κρατών μελών. Θεωρούμε ότι είναι αποφασιστική σημασίας. και στα πλαίσια της αλληλεγγύης πάντα και της συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε κύριε. Ο κύριος Δίνος Βρετός, πρόεδρος της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Ελλάδας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα της ε, συνεργασίας για το τόσο σοβαρό θέμα της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Η συνθήκη της Λισαβόνας αφορά την εφαρμογή του πρωτοκόλου 1 της συνθήκης ε, για τα εθνικά κοινοβούλια και τις δυνατότητες των κοινοβουλίων να συμμετέχουν στα θέματα κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Το σημαντικό γεγονός στη νέα συνθήκη είναι η δημιουργία του θεσμού του ύπατου εκπρόσωπου και της κάτω από αυτών Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αν και στα θέματα της ΚΕΠΑ, παραμένει ως αποφασιστικό σώμα η Επιτροπή Άμυνας που υπάγεται πλέον και αυτή στον ύπατο εκπρόσωπο. Σύμφωνα με τη συνθήκη, οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία και είναι αυτό που προσδιορίζει το διακυβερνητικό χαρακτήρα της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Από αυτό το διακυβερνητικό χαρακτήρα προσδιορίζεται και ο σημαντικός ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής. Ένα άλλο δεδομένο, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι μετά την κατάργηση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινοβουλευτική της συνέλευση, που ήταν το μοναδικό κοινοβουλευτικό όργανο που ασχολείται μέχρι τώρα με θέματα άμυνας, διακόπτει τις εργασίες της τον Ιούνιο του 2011. Είναι προφανές ότι στα πλαίσια της νέας συνθήκης πρέπει ως εθνικά κοινοβούλια να βρούμε το νέο μας βηματισμό. Υπάρχουν ήδη διαφορετικές σκέψεις και προτάσεις, ενώ στη διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων που θα γίνει τον Απρίλιο του 2011 αναμένεται να διαμορφωθεί και εκεί κάποια πρόταση. Όπως είπα, υπάρχουν ήδη προτάσεις που προέρχονται από το Γαλλικό και το Ιταλικό Κοινοβούλιο και τη Γερουσία. Και εκτιμώ ότι και άλλα κοινοβούλια θα διατυπώσουν τις απόψεις τους πολύ σύντομα. Είναι επίσης προφανές ότι η ανάγκη συνεργασίας των Ελληνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου ο ρόλος είναι προσδιορισμένος από τη συνθήκη, αλλά και από την πρόσφατη απόφαση της 16 Σεπτεμβρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι προσδιορισμένος και σίγουρα ε, είναι η βάση για τη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η άποψή μου, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι τα ελληνικά κοινοβούλια χρειάζονται μια συγκροτημένη και συστηματικοποιημένη αντιμετώπιση των θεμάτων τη κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Στα πλαίσια αυτά, ένα κοινό διακοινοβουλευτικό σώμα, στο οποίο θα μπορούσαν να, συμμετέχουν, να συμμετέχει και το Ευρωκοινοβούλιο, είναι εντελώ απαραίτητο. Δεν μιλάω για ένα νέο όργανο στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάω όμω για μια συγκροτημένη παρουσία των ειδικών κοινοβουλίων όπου θα έχουμε μια γραμματεία όχι μεγάλη αλλά μια γραμματεία επαρκή να στηρίζει αυτή τη λειτουργία. Θα πρέπει να έχουμε επιτροπές αντίστοιχες με εκείνες που αφορούν θέματα της κοινή ευρωπαϊκής ε, ε, αμυντικής και, αμυντικής ε, και πολιτικής ασφάλειας. Θα πρέπει να έχουμε εισηγητές και εκθέσεις για να μπορούμε να είμαστε ουσιαστικοί και υποβοηθητικοί του έργου των κυβερνήσεών μας. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, αρκετές αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Ε, υπάρχουν αντιδράσεις που προέρχονται από συναδέλφους μας ε, του, Εθνικού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και από ο άλλος καλοπροέδρες αντιδράσεις ότι δηλαδή μπορεί να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο σώμα, ότι μπορεί το κόστος να είναι μεγάλο, Όλα αυτά τα γνωστά. Τα έχουμε αντιμετωπίσει και σε άλλες περιπτώσεις. Όμως εγώ πιστεύω ότι το να έχουμε 5-6 άτομα να, στηρίξουν μια, να έχουμε μια γραμματική, γραμματιακή υποστήριξη από 5-6 άτομα δεν είναι τίποτα. Εδώ παίρνουμε, ασχολούνται με την νέα υπηρεσία εξωτερικής δράσης 5.000 άτομα. Είναι αστείο κατά την άποψή μου να λέμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα <laughs> από την λειτουργία 5-6 ατόμων για την γραμματιακή υποστήριξη ενός τέτοιου σώματος. Ε, πιστεύω ε, ότι και το, ε, το, έχω ακούσει και από τον κύριο Μπροκ χτες στα πλαίσια της συζήτησης που κάναμε στη Λισαβόνα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να στηρίξει αυτή τη λειτουργία με δική, της, δική του γραμματιακή υποστήριξη και μπορεί να ελέγχει κατά κάποιο τρόπο όλη αυτή την, την υπόθεση τα ελληνικά κοινοβούλια είναι ανεξάρτητοι φορείς. Και ο φορέας που θα λειτουργήσει για την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα πρέπει επίση να είναι ανεξάρτητο, Για να είναι αποτελεσματικό. Διαφορετικά δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο από το να συναντιόμαστε εδώ, άτυπα στην ουσία, χωρί να έχουμε καμία προετοιμασία, να χωρίς να έχουμε καμία έκθεση και κανέναν εισηγητή, να συζητάμε διάφορα θέματα και να φεύγουμε ικανοποιημένοι. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε δεν το έχουμε κάνει. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώντας σας για άλλη μια φορά που μου δίνετε την ευκαιρία, την ευκαιρία να εκφράσω την άποψή μου, προτείνω να σκεφτούμε το σημαντικό γεγονός μιας νέας συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά με βάση μια συγκροτημένη, ε, ένα, ένα συγκροτημένο σώμα το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βρετό. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή των συναδέλφων στο γεγονός ότι αυτό το πρώτο μέρος εργασιών ε, μετά την εισαγωγή του Υπουργού Σαστέλ αφορά την ενίσχυση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας όσον αφορά την νομιμότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δηλαδή την εισήγηση του κυρίου Ντανζάν, το δεύτερο μέρος δηλαδή της ημέρας μας, θα αφορά την ανάπτυξη αυτού του θέματος και μπορείτε να αναπτύξετε να προβάλλετε τη σκέψη σας τότε, αλλά για λόγους οργάνωσης θα ήταν σκόπιμο να αρκεστείτε σε αυτά τα δύο θέματα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη. Τώρα έχουμε την πρώτη παρέμβαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Άντριου Νταφ έχει το λόγο εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Κύριε Νταφ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τρία σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι να αξιολογήσουμε, να εκτιμήσουμε σωστά τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία της εθνικής στρατιωτικής δυναμικότητας, των εθνικών στρατιωτικών δυναμικοτήτων. Χρειάζεται γι' αυτό μια συστηματική ανάλυση κόστους οφέλους που θα διεξαχθεί στο σύνολο των 27 κρατών μελών μας ώστε να αξιολογήσουμε την ικανότητά μας να παρεμβαίνουμε, να ενεργούμε αποτελεσματικά και ουσιαστικά σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Προτού ολοκληρωθεί μια τέτοια ενδελεχής αξιολόγηση δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποια θα είναι τα μέτρα που θα χρειαστεί να λάβουμε για να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των στρατιωτικών μας δυνάμεων και την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ στρατιωτικού και πολιτικού σκέλους. Διότι αυτό, αυτά θα είναι μόνο εικασίες Χρειάζεται λοιπόν μια αξιολόγηση πάνω στην οποία θα στηρίξουμε τον μελλοντικό μας σχεδιασμό. Μια αξιολόγηση η οποία θα μας δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Κάτι που δεν διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Κάθριν Άστον πρέπει να προσδιορίσουν ένα χρονοδιάγραμμα για μια δομημένη και συνεχιζόμενη συνεργασία. μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτό είναι ένα θέμα σύνθετο και θα απαιτηθεί χρόνος προτού να μπορέσουμε να επιλέξουμε την οδό, τον δρόμο που θα χρειαστεί να ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα. Πρέπει να ληφθεί μια ουσιαστική απόφαση. για το κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να ενταχθεί στην κεντρική ομάδα των κρατών που διαθέτουν στρατιωτική ικανότητα. Και ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το εξής. Εάν δεν ε, προσδιοριστούν οι στρατηγικές μας σχέσεις με την Τουρκία, οποιαδήποτε ελπίδα ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ θα αποδειχθούν άσκοπες. Η πολιτική προτεραιότητα για την Κάθριν Άστον πρέπει να είναι λοιπόν η διευθέτηση του, της τουρκοκυπριακής, του, του Κυπριακού, συγγνώμη, του Κυπριακού. Ευχαριστώ κύριε Νταφ. Το λόγο τώρα έχει ένας ε, Ιταλός συνάδελφος, ο κύριος Εντμόντο Τσιριέλη, πρόεδρος της Επιτροπής Αμήνης ε, της Βουλής Ιταλίας. Ε, Ευχαριστώ. Καλημέρα Πρόεδρε, καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, ούτε να μπω σε λεπτομέρειες για τη σημασία των συνθήκων και τη συνθήκη τη Αβώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει την ολοκλήρωση και τη συμπροματικότητα της πολιτική και της στρατιωτική δράση με το ΝΑΤΟ. Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συνεργασία και να επαναληφθεί η συνεργασία με τη Ρωσία γιατί είναι στρατηγικού ενδιαφέροντος νομίζω για την Ένωση η Ρωσία να ε, συμμετέχει πλήρως στις δράσεις σταθεροποίησης και ειρήνευσης στον κόσμο γιατί βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας μεγάλος γείτον της ε, Ένωσης. Και θα ήθελα να καλέσω ε, όλους τους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγαλύτερη αλληλεγγύη ε, ως προς το Αφγανιστάν και στην παρέμβασή μας εκεί. Σήμερα αρμόζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλη προσπάθεια και οικονομική αλλά όχι μόνο. Η Ιταλία σήμερα 2 δισεκατομμύρια ευρώ πληρώνει το χρόνο για την αποστολή στο Αφγανιστάν. Πέρα από το τεράστιο ανθρώπινο κόστος, καταλαβαίνετε, διότι ε, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, η παρέμβαση είναι προτεραιότητας για την ασφάλεια στον κόσμο και ε, συνεπώς και για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη στο βαθμό των δυνατοτήτων τους να ε, συμμετέχουν με τρόπο πιο αλληλέγγυο. Σε ό,τι αφορά την αμυντική βιομηχανία, άλλο στρατηγικό θέμα τώρα για την ΕΠΑ στην Ευρώπη, θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, την ολοκληρωσή μα, τη συνεργασία μας ε, και να εφαρμοστούν πλήρω οι δύο οδηγίε Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τη μείωση τη γραφειοκρατία και τι εξαγωγέ. Και επίση θα πρέπει να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό ε, όσο αφορά την παραγωγή αλλά και την έρευνα. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και αν ε, ε, δίνει λιγότερα χρήματα από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχει 89 προγράμματα ε, ερευνητικά. Κατακαιρματίζεται αυτή η προσπάθεια, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε κάτω από 30. Για τις ένοπλες δυνάμεις επίσης χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία και ολοκλήρωση και μέσω ε, κοινών ασκήσεων, ανταλλαγών, ε, ενημέρωσης και στις ε, στρατιωτικές σχολές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πιο συγκεκριμένη και είναι απαραίτητο να μορφώνεται καλά το στρατιωτικό μας προσωπικό πάντα για την κοινή προσπάθειά μας. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και τέλος, σημειώνουμε ε, αυτό που γίνεται μετά τη διάλυση της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν κοινέ ε, συνεδριάσεις εργασίας τύπου της σημερινής, αλλά ίσως θα μπορούσε να συμμετέχει εκεί και η κυρία Άστον για να δείξει ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια συμμετέχουν και συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Τώρα δίνουμε το λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον κύριο Κρίστιαν Χέλλερ. Από το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αφαιρθώ σύντομα στον τομέα της στρατιωτικοπολιτικής συνεργασίας. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναλάβουμε δράση εδώ και ο πρόεδρος Ντονζόν της ε, Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας το προώθησε πάρα πολύ. Στο θέμα αυτό της στρατιωτικής πολιτικής συνεργασίας είναι ένας τομέας που πιστεύουμε ότι πολύ γρήγορα, πολύ πρακτικά μπορεί να εμφανίσει μια εμβάθυνση της ευρωπαϊκής προσπάθειας. Χαίρομαι που παρευρίσκεται και η κυρία Νό εδώ που κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό και στο μέλλον για τον τομέα αυτό και χαιρόμαστε και τονίζουμε ακριβώς που θέλετε να εντείνετε τις προσπάθειές σας και ε, επίπεδο είπα τη εκπροσώπου. Γιατί το λέω αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν και οι φίλοι από τα εθνικά κοινοβούλια ότι το Συμβούλιο ε, είχε ορίσει από πέρυσι κάποιες δομές που πολιτικά έχουν ολοκληρωθεί και έχει δώσει και τις ευλογίες του. Με 11.000 λοιπόν ε, προσωπικό θα πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον τρεις δράσεις, στρατιωτικοπολιτικές, πολιετής με διαφορετική ένταση κάθε φορά, ε, άλλοτε περισσότερο πολιτική, άλλοτε περισσότερο στρατιωτική. Τώρα, η πραγματικότητα ποια είναι στην Ευρώπη ότι έχουμε περίπου 3.000 ε, ε, άνδρες στις αποστολές μας, κυρίως πολιτικού περιεχομένου και έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες στην ανάπτυξη του προσωπικού εκεί και στην ε, ασφάλειά του. Γι' αυτό αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην τα συζητάει αυτά έτσι με μεταφυσικό και θεωρητικό τρόπο, αλλά από τα θεμέλια των όσων ήδη έχουμε αποφασίσει. Τι ισχύει, τι είναι λειτουργικό, τι είναι επιχειρησιακό, ποιε είναι οι πραγματικότητε επιτόπου και οι δομικέ. Και θα πρέπει να πούμε ότι οι εθνικέ κυβερνήσει, στο σχεδιασμό που κάνουν και στου στόχου αλλά και στι αποφάσει του, είναι πολύ πιο μπροστά από την πραγματικότητα ε, και θα πρέπει ας πούμε, να προσγειωθούμε στη σημερινή κατάσταση που διαμορφώνουμε συγγνώμη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και βλέπουμε και τις επιχειρησιακές δομές και τη λειτουργία, θα πρέπει να ασχοληθούμε για πρώτη φορά ε, με το να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτά τα πράγματα. Και επίση και τα κράτη-μέλη, και πολύ σημαντικό για του εθνικού βουλευτέ, τα κράτη-μέλη λοιπόν, που έχουν αποφασίσει κάποια πράγματα πολύ μακρόπνοα, ε, δεν είναι του παρόντος. Θα πρέπει να κλείσει αυτό το χάσμα, γιατί οι εξελίξεις δεν ακολουθούν. Ας φανταστούμε ότι είχαμε μια δεύτερη αιτία αυτή τη στιγμή, μια μεγάλη θεομηνία τέτοιας διαστάσεως, με την ανάγκη ακριβώς να στείλουμε και στρατιωτικές εκεί δομές. Ως Ευρώπη σήμερα δεν θα ήμασταν σε θέση να ανταποκριθούμε ε, στις υποχρεώσεις που ήδη έχουμε επιβάλει στους εαυτού μας. Και το πρόβλημα αυτό είναι και πολιτικό και πρόβλημα αξιοπιστία για την ευρωπαϊκή κοινότητα αλλά και για τα κράτη-μέλη. Και διεθνώ μα εκθέτει. Ε, γι' αυτό αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εστιάσουμε ε, πολύ συγκεκριμένα πώ μπορούμε να αναπτύξουμε την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε άλλε αποφάσει όχι. Να δημιουργήσουμε τι δομέ συγκεκριμένα. Γι' αυτό έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για το διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί έχουμε λίγο την αίσθηση ότι οι κυβερνήσει πώς να το πω, έχουν λάβει κάποιες αποφάσεις τις οποίες τώρα για λόγους πολιτικούς, οικονομικούς, διαρθρωτικούς, ξέρω εγώ, βλέπουμε ότι στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν οι λιμένες, επαναλαμβάνω, αποφάσεις. Και ένα τελευταίο, σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό σκέλος. Και πάλι ας μην προσανατολιζόμαστε σε πολιτικά θέματα. Έχουμε ε, τις, ε, τους μάχημους σχηματισμούς, τα λεγόμενα battle groups. Από τη χρηματοδότηση όμως τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι μόνο το Nordic Battle Group που υποτίθεται ότι έχει διαλυθεί αλλά από τις βορειοευρωπαϊκές ευρωπαικες χώρες που έχουν συνεισφέρει στη ε, συγκέντρωσή του έχει φτάσει σε μια κατάσταση που λέει έχουμε αποκομίσει εμπειρίες, έχουμε φτιάξει δομές και στο μέλλον θα μπορούσαμε να το επανασυστήσουμε αυτό το, το σχηματισμό. Ενώ όλοι οι άλλοι σχηματισμοί διαλύονται και δεν έχουν και καμία ουσιαστική επιρροή στο μέλλον. Λοιπόν, και αυτό να το σκεφτούμε. Πώς να ε, συνδυαστεί καλύτερα ο πολιτικός και ο ε, στρατιωτικός σχεδιασμός. Έχει νόημα να φτιάχνουμε μάχημους σχηματισμούς, να τους χρησιμοποιούμε, μετά να τους διαλύουμε και στη συνέχεια τι. Τώρα και ένα μηχανισμό στρατιωτικό των Αθηνών, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ε, και πώς θα το λέμε, αλλά να μην επιβαρύνει ε, και το κόστος λειτουργίας του μάχημου ε, σχηματισμού αποκλειστικά και μόνο το κράτος που ήταν υπεύθυνο κάποια χρονική στιγμή για τη σύστασή του. Αυτό είναι και εις βάρος των μικρών κρατών, καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χέλλερ. Δίνουμε το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της ε, Βουλής των Αντιπροσώπων της ε, Λιθουανίας. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε. Αυτή είναι η πρώτη συνεδρίαση τη σημερινή μας συνάντησης που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική και θα έπρεπε να ανατρέξουμε στη γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ιδέες και στις σκέψεις ε, του Ρομπέρ Σουμάν. Εάν λοιπόν επιστρέψουμε στις ρίζες, βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκαν 10 μετακομμουνιστικές χώρες μετά από κάποιο διάστημα και για μας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση δημοκρατικών κρατών. 27 στο σύνολό τους. Όλοι, όλοι έχουμε την ίδια ε, στάση και την ίδια προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές και αξίες. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε εστιαζόμαστε στην μελλοντική πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν συζητάμε για τέτοια θέματα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη στα άλλα κράτη ανά τον κόσμο που συμμερίζονται τις ίδιες αξίες και αρχές με εμά. Έχοντας κατά νου ότι δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε τις ε, δραστηριότητες και τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ. Η συνεργασία με, την Ευρωπαϊκή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για την χώρες της Κεντρικής Ευρώπης στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου οι ε, Ηνωμένες έπαιξαν σημαντικό ρόλο εξασφαλίζοντας το δημοκρατικό μας μέλλον και επιτρέποντάς μας να ξεπεράσουμε 50 χρόνια σκλαβιάς, δουλείας. Πιστεύουμε λοιπόν όμως παρόλα τα αυτά ότι δεν πρέπει να υπάρχει διπλοποίηση των δράσεων και των δομών. Και υπάρχουν, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αφορά την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ας θυμηθούμε το ρόλο μας στην Ουκρανία. Ο ρόλος μας ε, υπήρξε πολιτικός σε αυτές τις χώρες. Θελήσαμε να παίξουμε ρόλο διαμεσολαβητή στα σύνορα. Η υπερδυνιστερία, η οποία είναι γεμάτη από στρατό, από στρατεύματα, απειλεί τη σταθερότητα στη Μολδαβία. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να, να είχαμε λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Ε, ελπίζω ότι θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στον αγώνα μας κατά της πειρατείας ε, από ό,τι άλλες μας ε, προσπάθειες στο παρελθόν. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η υπηρεσία της Βαρόνης Άστον πλαισιώνεται από εκπροσώπους των Υπουργείων Εξωτερικών. Αλλά ίσως ε, θα έπρεπε να γίνει ε, κάτι ανάλογο με το Υπουργείο Άμυνας, δηλαδή να υπάρχουν και εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας σε αυτή την υπηρεσία. Είναι κάτι που το σκεφτόμαστε στη Λιθουανία. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το στρατιωτικό σκέλος στην υπηρεσία της Βαρόνης Άστον. Ωστόσο θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις για την απόσπαση ε, ε, υπαλλήλων από ε, το Υπουργείο Άμυνας στην υπηρεσία της. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Κύριε Πρόεδρε, Χαίρομαι για αυτή την ευκαιρία διαλόγου με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι είναι ύψης της σημασίας για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, καθώς και την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αρμόζει σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό ακριβώς δημιουργήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η πολιτική μας στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και της άμυνας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβει η κυρία Άστον ένα μήνυμα και, τα, και από τα Εθνικά Κοινοβούλια έτσι ώστε να συμμετέχουν και τα δύο ε, φύλλα εξίσου, να υπάρχει ισότητα εκπροσώπησης των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Μέσα στα πλαίσια του οπλοστασίου μας θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα στρατιωτικής και πολιτικής ικανότητας, ιδιαίτερα στις ε, παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως απορρέει από τις διάφορες αποστολές μας εδώ και πολλά χρόνια. Δεν πρόκειται για ε, μία διπλή αποστολή. Δηλαδή ακολουθούμε τη δομή του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ εξελίσσεται διαφορετικά μέσα στα πλαίσια μιας εκπόνησης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας στρατηγικής. Νομίζω λοιπόν ότι προβάλλουμε μια εταιρική σχέση μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ με τις ΗΠΑ. Και γι' αυτό εμείς θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας στον ε, τομέα συνεργασίας με το ΝΑΤΟ και για την άμυνα και την ασφάλεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε περισσότερο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια των ε, μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους στόχους μας. Αυτή είναι μία ευκαιρία σε ευρωπαϊκό πλαίσιο για να παρέμβουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε πολλές παρεμβάσεις είτε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ είτε ε, εξιδίων. Θα πρέπει να παρέμβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι πολλές φορές και το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να φτάσει σε κρίσιμες ε, και επίμαχες περιοχές του κόσμου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξορθολογήσουν τη χρηματοδότηση στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας θα πρέπει να ορίσουμε τους εξοπλισμούς που χρειαζόμαστε και όπως ελέγχθη θα πρέπει να συνεννοηθούμε με τις βιομηχανίες άμυνας και να προωθήσουμε μία κοινή πολιτική στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Το Startup Fund το οποίο ε, δημιουργήθηκε και προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν αρκεί. Θα πρέπει να βρούμε άλλα μέσα για να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη να παρέμβουν και με ένοπλες δυνάμεις, με στρατιωτικές δυνάμεις. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας είναι πολύ σημαντική υποστήριξη και χρειαζόμαστε βεβαίως και την υποστήριξη Τη της ύπα εκπροσώπου. Ε, δεν θα πρέπει να μας διακατέχουν οι, οι του Βρετανικού establishment όπως ε, ίσχυε στο παρελθόν. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτήν την καθεστική τάξη και πιστεύω ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό το σκεπτικό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η διάρθρωση θα πρέπει να συνεχιστεί συνεχείς επαφές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτό και η κυρία Άστον, ιδιαίτερα στο θέμα της ασφάλειας στο, στην περιοχή του Σαχέλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαδραματίσουμε το ρόλο που μας ε, αρμόζει και όπως είπε και ο Άντριου Νταφ, υπάρχουν θέματα που θα πρέπει να επιληθούν εξ ολοκλήρου, διότι δεν πρόκειται για θέμα διένεξης έθνης μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου. Το θέμα είναι ευρωπαϊκής εμβέλειας και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί για να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τις διαφορές και σε άλλα μέρη του κόσμου. Δηλαδή, Πώς ε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό αν δεν μπορούμε να επιλύσουμε μια διαφορά μεταξύ της Κύπρου και μιας υποψήφιας χώρας για προσχώρηση. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή από τα Εθνικά Κοινοβούλια, θα ήθελα να σας δώσω ορισμένες ε, οργανωτικές πληροφορίες. Ξέρω ότι γνωρίζετε ότι αρχίζει απεργία των αερογραμμών σήμερα το απόγευμα. Άρα όσοι πρέπει να επιστρέψετε σήμερα θα πρέπει να δείτε αν μπορείτε. Η γραμματεία πληροφορείται, λαμβάνει πληροφορίες γιατί μάλλον είναι προειδοποίηση απεργίας, δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί και πριν από το τέλος του πρωινού θα σας δώσουμε ε, πληροφορίες ο κύριος Φρουνζούλικα από, το, ε, από τη Ρουμανική Βουλή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ μεταξύ ημών για να συζητήσω για ένα τόσο σημαντικό θέμα που είναι η ΕΠΑ καθώς και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, έχουν γίνει πολλές μελέτες που αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οικονομικός και κοινωνικός γίγαντας, αλλά δυστυχώς είναι ένας νάνος όσον αφορά την πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Και γι' αυτό έχω και ένα ερώτημα προς την ύπατη εκπρόσωπο προς τη Βαρόνη Άστον που είναι παρούσα σήμερα εδώ και νομίζω ε, ότι τουλάχιστον μία επόμενη φορά, με συγχωρείτε λέει ο μιλητής, έκανα λάθος, επειδή δεν βρίσκεται σήμερα εδώ, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τη συναντήσουμε κάποια άλλη φορά θα πρέπει να μας ε, απασχολήσει ε, η ρήτρα επίθεσης. Η ρήτρα επίθεσης όπως απορρέει από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αναφερόμαστε στο άρθρο 51 της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας και σε περίπτωση επίθεσης κατά ενός κράτους μέλους. Αυτή η ρήτρα ανταποκρίνεται στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ αναφέρομαι στο άρθρο 5 της Συνθήκης των Βρυξελών όπως τροποποιήθηκε και όπως έχει μεταφερθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών και αναφέρομαι στα 21 κράτη-μέλη που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ θα ασχοληθούν με τη συλλογική άμυνα και ασφάλεια μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αλλά θα ήθελα να προβάλλω ένα ερώτημα προς την ύπατη εκπρόσωπο, τη Βαρόνη Άστον. Πώς θα ισχύσει αυτό το άρθρο αμοιβαίας αρρωγής σε περίπτωση εναντίωσης ή επίθεσης κατά κράτους μέλος που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και εδώ μιλάμε για μια ευαίσθητη ζώνη στα πλαίσια της άμυνας και ασφάλειας. Δηλαδή τι θα γίνει πέρα από τα 21 κράτη-μέλη που συμμετέχουν και στο ΝΑΤΟ και στις δομές του ΝΑΤΟ πώς θα ανταποκριθεί η ύπατη εκπρόσωπος σε αυτή τη συλλογική άμυνα και ασφάλεια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Φρουντζούλικα. Το λόγο έχει ο κύριος Αρναούτ από την Πορτογαλική Βουλή. Θα ήθελα Καταρχήν να σας ε, ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή. Πιστεύω ότι πρόκειται για μία κοινή ε, προσπάθεια που επιτρέπει τη συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων και πιστεύω ότι το θέμα είναι άκρος επίκαιρο. Θα ήθελα να τονίσω ότι ε, δεν μας ενδιαφέρει, μάλλον δεν ενδιαφέρει μόνον η παγιοποίηση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Θα πρέπει να έχουμε λειτουργικούς μηχανισμούς και ένοπλες δυνάμεις που να είναι καλώς εξοπλισμένες και να προβάλλουμε μια ευρωπαϊκή βιομηχανία άμυνας που να έχει παγκόσμια εμβέλεια. Ζούμε μια εποχή κρίσης και όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες. Έχουν δηλαδή να αντιμετωπίσουν άλλα θέματα, άλλες προτεραιότητες Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε το ρόλο της άμυνας, διότι και εδώ διανύουμε μια κρίσιμη κατάσταση και σε αυτό το τομέα. Γίνονται πολλές επενδύσεις και δαπάνες και δαπανάτε ένα 2% του ΑΕΠ, ίσως και λιγότερο από πολλά κράτη-μέλη, για δαπάνες άμυνας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο διαφέρει από τις διεθνείς επιταγές δαπανών στον τομέα της άμυνας. Υπάρχουν και αναδυόμενες χώρες όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία και οι χώρες της Μέσης Ανατολής όπου οι επενδύσεις άμυνας είναι αστρονομικές και ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας νέας ισορροπίας διεθνώς. Γι' αυτό θα πρέπει να συντονίσουμε την δράση των ενόπλων δυνάμεων για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ΕΠΑ. θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν το κάνουμε αυτό, ίσως διαθέτουμε τους καλύτερους μηχανισμούς συντονισμού στην άμυνα και ασφάλεια, αλλά θα αποδυναμώνεται ο ρόλος μας ως προς δράσεις διεθνούς εμβέλειας, αν δεν έχουμε καλούς εξοπλισμούς και ένα δυναμικό ασφάλειας το οποίο να είναι καλώς εξοπλισμένο έτσι ώστε να μπορεί να δρά συντονισμένα και με ευελιξία. Επίσης, εάν θέλουμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο, γενικότερα, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να υποβοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Άμυνας, διότι θα χάσουμε τον προεξάρχοντα ρόλο μας. Υπάρχουν δύο μέσα. Ένοπλες δυνάμεις και δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας που να είναι καλώς εξοπλισμένες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες εχμής για να μπορέσουμε να δράσουμε στο διεθνές προσκήνιο με τον καλύτερο δυνατό συντονισμό. Διαφορετικά θα αποδυναμωθούμε. Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες της ΕΠΑ. Χωρίς αυτούς τους δύο πυλώνες δεν θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρώπης στο διεθνές προσκήνιο. Γι' αυτό θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα πρέπει να την χάνει ενδελεχούς ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης να δημιουργηθούν και εθνικοί μηχανισμοί για αυτή την εποπτεία. Δεν χρειάζεται μόνο συντονισμός. Πρέπει να δράσουμε ενεργά και να έχουμε ένοπλες δυνάμεις που να είναι ε, παρούσες στο διεθνές προσκήνιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αρναούτ. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρέμβει ο κύριο Τάνοκ που είναι συντονιστής της ομάδας, της, της, του, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το κόμμα μου, η Βρετανή Συντηρητική στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική για την ΚΕΠΑ ή την ΕΠΑ διότι υπήρχε κίνδυνο, στον τον οποίο αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι, τη αποσύνδεση από τι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής που παραμένουν η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο και η υπονόμευση του ΝΑΤΟ που μας εγγυάται ασφάλεια και ειρήνη για τόσο πολύ μεγάλο διάστημα στην Ήπειρό μας, καθώς και διπλοποίηση των προσπαθειών του ΝΑΤΟ, όταν τα αμυντικά μέσα είναι ήδη τόσο περιορισμένα στις σημερινές συνθήκες λιτότητας που γνωρίζουν όλες οι χώρες μας και οι περικοπές στους αμυντικούς προϋπολογισμούς. Στον Ηνωμένο Βασίλειο μάλιστα αυτή τη στιγμή γίνεται μια επανεξέταση ε, των αμυντικών δαπανών που ασφαλώς θα καταλήξει σε περικοπές αυτών των δαπανών. Και νομίζω ότι όλοι θα παραδεχθούν ότι οι δυνάμεις μας είναι πάρα πολύ καλές και απαραίτητες για τις δράσεις στο Αφγανιστάν και οποιαδήποτε μείωσή τους θα επηρεάσει σημαντικά τη σταθερότητα παραδείγματο χάρη στο Πακιστάν. Γι' αυτό λοιπόν στα πλαίσια της ΕΠΑ πρέπει να συντονίσουμε τις δράσεις μας με εκείνες του ΝΑΤΟ. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνάλληση του ΝΑΤΟ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχω παρατηρήσει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τους τελευταίους μήνες ότι ε, μεταξύ των αξιωματούχων του ΝΑΤΟ και στη συνέλευση και μεταξύ των βουλευτών από τις διάφορες χώρες υπάρχει πλέον αποφασιστικότητα και δέσμευση για απτά και ικανοποιητικά αποτελέσματα Επιτροπή μας ε, ε, άκουσε πρόσφατα τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ρασμούντσεν, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, ενώ αποτελεί πλέον μια συνήθη διαδικασία συμμετέχουμε επίση τα, ε, κοινοβούλια, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλίων συμμετέχουν ενεργά στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο συνασπισμός στη, στη, η κυβέρνηση συνασπισμού στη χώρα μου έχει αλλάξει στάση σε σχέση με την ΕΠΑ. αναγνωρίζοντας τις δράσεις στο κέρας της Αφρικής και κατά της πειρατείας στα ανοιχτά της Σομαλίας, μιας ιδιαίτερα ευάλωτης χώρας αυτό που διδάχθηκα ως μέλος Υποεπιτροπής Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι χώρες όπως η Ινδία και συμμετέχουν αντιπροσωπεία της Ινδία είναι πλέον διατεθειμένες να συνεργαστούν με τις ε, ε, δυνάμεις της ΕΠΑ ενώ ένα ΝΑΤΟ το οποίο ε, ε, στο οποίο ε, κυριαρχεί, στο οποίο επικρατούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, για μια τέτοια συνεργασία υπάρχουν από πολλέ χώρες πολύ πιο ουσιαστική δισταγμή. Και έχω σημειώσει συχνά ότι σε κοινοβούλια όπου επικρατούν οι σοσιαλιστές είναι πιο, καλύτερα ε, γίνεται πιο αποδεκτό το να συμμετέχει κάποιος σε μια δράση που διεξάγεται από την ΠΑ παρά σε μια δράση στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τους επόμενους μήνες μέχρι το Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να υποστηρίξει τις ε, ε, συνομιλίες στην Κύπρο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών διότι τα εμπόδια που δημιουργεί διαρκώς η Τουρκία ε, είναι μια κατάσταση πλέον που δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί. Εάν λοιπόν ξεπεράσουμε τα προβλήματα και έχουμε μία, ε, πλέον μία Κύπρος που θα είναι ένα νέο κράτος κάτω από μία σημαία, αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και αν μπορεί ε, κάτι να κάνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σημαντικό. Θα εγγενιαστεί μια έκθεση σήμερα το απόγευμα για τα διάφορα πρόσωπα της Κύπρου και σας παρα προσκαλώ να έρθετε να ρίξετε μια ματιά σε αυτή την έκθεση. Εγώ είμαι βουλευτής ε, για το Λονδίνο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι, έχει πλέον αναλάβει πλή, πλήρη δέσμευση, είναι προσιλωμένο στην προώθηση τη ΕΠΑ. Ευχαριστώ για την προσοχή Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Ολοκληρώνει τη συζήτηση ο κύριος Αβέροφ Νεοφίτου τώρα που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Βολής των Αντιπροσώπων της Κύπρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γνωστό ότι όσο και αν συζητούμε στο να βρούμε τους καλύτερους τρόπους συνεργασίας Ευρωκοινοβουλίου, Επιτροπής, μαζί με την κυρία Άστον ή ακόμα και Εθνικών Κοινοβουλίων, ποτέ δεν θα πετύχουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη και αξιόπιστη εξωτερική πολιτική. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουν 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί εξωτερικών ζητημάτων να μιλούν με μια φωνή. Αλλά και αυτό δεν είναι αρκετό αν δεν υποστηριχτεί με μια αξιόπιστη άμυνα και πολιτική ασφάλειας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα ήθελα κλείνοντας κύριε Πρόεδρε να κάνω και ένα σχόλιο και να συμφωνήσω με κάποια ζητήματα που έχουν εγερθεί από συναδέλφους βουλευτές και ευρωβουλευτές ότι πρέπει να επιληθεί το κυπριακό ε, και όλοι πρέπει να συμβάλλουμε και η Κύπρος είναι η τελευταία που θα ήθελε να δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Καταβάλουμε προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού για να ξεπεραστούν και τα προβλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Και θα ήταν καλό ε, και η Τουρκία να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Νεοφίτου. Πριν δώσουμε το λόγο για να απαντήσει και να ολοκληρώσει ο κύριος Υφυπουργό, ε, να σας πω ε, ειδήσει νέα που έχουμε για την απεργία, ε, την επαπειλούμενη. Μαθαίνουμε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των συνδικάτων και των αρχών του αεροδρομίου. Δεν ξέρουμε ακόμα την έκβασή τους στις 12 θα βγει ανακοίνωση και θα σας ενημερώσουμε για να μπορέσετε να κανονίσετε την πορεία σας και να έχετε και κάποιες ενδείξεις για την οργάνωση της επιστροφής σας. Να ξέρουμε τη διάρκεια, την εμβέλεια, την έναρξη και γενικά περισσότερες λεπτομέρειες για την προβλεπόμενη απεργία. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τα ε, πιο σημαντικά θέματα εξωτερική πολιτική που ακούσαμε. Κύριο Σαστέλ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σα πω ότι συζήτησαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θα δοθεί και συνέχεια οπωσδήποτε από πλευράς κυρία Άστον τη ίδια Έχει ε, προγραμματιστεί η παρέμβασή της ε, στο Κοινοβούλιο στις 27 Οκτωβρίου και στη διάσκεψη των Προέδρων και στην Επιτροπή Εξωτερικών στις 18 Οκτωβρίου. Επιτρέψτε μου να δώσω μερικές απαντήσεις τώρα. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ρήτρα αλληλεγγύης, η αμοιβαία συνδρομή. Ε, αναφερθήκατε πολύ σε αυτή. Υποχρεώνει η ρήτρα αυτή τα κράτη-μέλη και την Ένωση να ε, βοηθούν μια χώρα όταν υφίσταται τρομοκρατική επίθεση, θεομηνία, ανθρωπογενή καταστροφή και με στρατιωτικά μέσα. Αυτή η ρήτρα γνωρίζετε επίσης ότι δεν έχει σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Είναι σημαντική διάταξη μεν, αλλά και πάρα πολύ περίπλοκη, γιατί μπαίνουν πολλά στοιχεία εκεί. Πολιτική προστασία, ε, δικαιοσύνη, εσωτερικά θέματα, καταπολέμηση της θερμοκρατίας και εφαρμογή της απαιτεί συγκεκριμένη και κοινή πρόταση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο. Και ε, σε ό,τι αφορά την προσφυγή σε στρατιωτικά μέσα, ε, να στην κυρία Άστο να κάνει εκείνες τις προτάσεις που θεωρεί κατάλληλες. Δεν χρειάζεται να θυμίσω ότι ήδη έχουμε ένα μηχανισμό υποστήριξη σε περίπτωση εσωτερικών κρίσεων, όπω το κέντρο παρακολούθηση και ενημέρωση, στο οποίο τα κράτη-μέλη μπορούν να, απευθυνθούν για να ζητήσουν βοήθεια και συντονισμό σε περίπτωση κρίσης. Είναι στο Συμβούλιο αυτή η υπηρεσία. Τώρα, αναφερθήκατε στην ενίσχυση του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού ελέγχου στα πλαίσια ε, της ε, ΕΠΑ. Η ύπατη εκπρόσωπος έχει κάνει μια ανακοίνωση και δήλωση για την πολιτική ευθύνη και ανακοίνωση και δεσμεύσεις από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ε, επικεφαλής ε, των αποστολών που διοικούν υψηλόβαθμού ε, ε, υπαλλήλου, έρχονται στο Κοινοβούλιο και ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ε, για τις εξελίξεις και τα πράγματα και στην ΕΠΑ. Και δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η άμυνα ιδιαίτερα είναι εθνική αρμοδιότητα και είναι ένα θέμα ευαίσθητο και λεπτό για τις κυβερνήσεις και συνεπώς για τα εθνικά κοινοβούλια. Βάση λοιπόν παραμένει η διάταξη του Συμβουλίου του, της Σύνθηκης που έχουν εγκρίνει και κυρώσει τα κράτη-μέλη και η δήλωση παριθμών 14 που λέγει ότι δεν εκχωρείται καμία νέα εξουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα στην πολιτική ε, ασφάλεια, στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, σε ό,τι αφορά τη διακοινοβουλευτική συνεργασία, σε εσά εναπόκειται, στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αποφασίσετε πώ θα διαμορφώσετε αυτή τη συνεργασία σα. σε ό,τι αφορά την ε, ανάληψη αποστολών και καθηκόντων από μικρές ομάδες κρατών μελών. Είναι γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε βαθύνει στη συζήτηση αυτή, όπως και στο μόνιμο διορθωτικό συντονισμό και συνεργασία χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή ε, της ΕΠΑ, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, αλλά η μόνιμη διαφθορτική συνεργασία δεν απαιτεί πάντα επίσημες αποφάσεις ε, για την εφαρμογή της. Βεβαίως η εφαρμογή μπορεί να γίνει μόνο βάση μιας αμοιβαίας και σαφούς αντίληψης για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Κατά τη διάρκεια της διαχείρισης κρίσεων, πώς μπορούμε λέτε να βεβαιωθούμε ότι τα στρατιωτικά στοιχεία δεν ε, κυριαρχούν. Από πλευράς ε, θεσμικής η πολιτική αυτή η ΕΠΑ έχει πολιτικό διοικητή και τα πολιτικά και τα στρατιωτικά στοιχεία και πτυχές υπόκεινται στην ε, ύπατη εκπρόσωπο και η πολιτική Επιτροπή Ασφάλειας εξασφαλίζει τη στρατηγική παρακολούθηση και των στρατιωτικών και των πολιτικών πτυχών και βασική πρόκληση είναι να έχουμε μια συνολική συνοχή προς τα έξω στη δράση μας λαμβάνοντας πάντα τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου. Η πολιτική διαχείριση των κρίσεων εντάσσεται σε ένα διευρυμένο τέτοιο πλαίσιο και βέβαια χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Έχει γίνει ιδέα μεγάλη πρόοδος στις συνέργειες ε, στη στρατηγική ε, για ένα σχεδιασμό ολοκληρωμένο πολιτικών και ε, στρατιωτικών πτυχών. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούν να βελτιωθούν οι δομές διοίκησης στο επιχειρησιακό επίπεδο και τέλος να βεβαιωθούμε πάντα ότι θα υπάρχει συνέργεια και ε, συμπληρωματικότητα του πολιτικού με το στρατιωτικό σκέλος και με ε, πραγματογνωμοσύνη με μελέτες και στα δύο σκέλη αυτά. Όπως είπατε και εσείς, ε, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα πρέπει να έχουμε όλη την εμπειρία και όχι μόνο διπλωμάτες και μια ισορροπία φίλου βεβαίως ανδρών και γυναικών. Γνωρίζετε ότι η κυρία Κάθρια Άστον είναι πάρα πολύ στρατευμένη σε αυτή την υπόθεση και στα πλαίσια της εφαρμογής του ψηφίσματος 1325 των Ηνωμένων Εθνών. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόοδο που έχει γίνει στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Η πρώτη φάση είναι η φάση της ε, συγκέντρωσης απόψεων για να καταλήξουμε σε μια κοινή αντίληψη. Γι' αυτό έγιναν δύο σεμινάρια με εκπροσώπους των κρατών μελών. Το τελευταίο μάλιστα ε, ήταν ε, βελγικής διοργάνωσης θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, αυτή την προσπάθεια για να συγκλίνουν οι απόψεις μας για θέσεις και διατάξεις πάρα πολύ συγκεκριμένες στις συνθήκες ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή και το καθορισμό των κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούνται. Ένα από τα σημεία στα οποία υπάρχει συνένεση είναι ότι η διαρθρωμένη συνεργασία, η μόνιμη αυτή, θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν, ε, χωρίς να αποκλείει κανέναν το θέμα τώρα που τίστε είναι πώς θα μπορούσε έτσι να βοηθήσει τη συνεργασία συγκεκριμένα νέα με τρόπο που ε, να δέχονται όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αμήνης έχει επιφορτιστεί με το έργο να κάνει περιοδική ε, ανάλυση των κρατών που συμμετέχουν ως προς τις ικανότητες τους και τις δυνατότητες και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχει από τη συνθήκη θα συνεχίσει αυτός ο οργανισμός να συντονίζει, να βοηθάει και να ε, συμπαραστέκεται στα κράτη-μέλη. Δύο λόγια σε ό,τι αφορά τώρα τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομής. Τα κράτη-μέλη υπόσχονται το ένα στο άλλο να συνδράμουν το ένα το άλλο σε περίπτωση ένοπλης εισβολής ή επίθεσης. Ε, έρχεται να συμπληρώσει την πολιτική συνεργασία στην άμυνα. Είναι πολιτική και νομική συνεργασία και θα μπορεί κανείς να προσφεύγει σε περίπτωση ανάγκης. Ωστόσο, η ρήτρα αυτή αμοιβαία συνδρομής προβλέπει ε, πιο δραστήρια εφαρμογή και θυμίζουμε ότι το ΝΑΤΟ είναι κάτι που ε, εγγυάται την άμυνα των μελών του και επίσης η συνθήκη αναφέρεται ρητά σε χώρες που έχουν παράδοση ουδετερότητας ε, μεταξύ των κρατών μελών. Πάνω σε αυτή η ρήτρα μεταθέτει το βάρος περισσότερο στα κράτη-μέλη τα ίδια και λιγότερο στο Συμβούλιο Υπουργών. Σε ό,τι αφορά τις δομές διοίκησης τώρα. Ε, και αυτό είναι ένα θέμα περίπλοκο όσο και σημαντικό για το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δρά και να αναλαμβάνει τις ευθύνες προστασίας των στρατιωτικών και των ε, αστυνομικών ε, πυρογνωμών ε, των κρατών μέλων. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει μια σειρά μηχανισμών ήδη για να γίνεται ο επιχειρησιακό σχεδιασμός και οι αποστολέ στην πράξη. Και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές αποστολέ, ο σχεδιασμό γίνεται από πολιτικούς, ενώ για τα στρατιωτικά έχουμε μηχανισμούς ε, που ε, προβλέπουν να συστήνεται ένα γενικό επιτελείο αυτή τη στιγμή, λαμβάνεται μια απόφαση για μια στρατιωτική αποστολή. Το θέμα είναι κατά πόσο οι σημερινοί μηχανισμοί θα ανταποκριθούν πλήρω στι ανάγκε μα. Γιατί αυτοί βασίζονται κυρίω σε εξωτερικέ ικανότητε που δραστηριοποιούνται, ενεργοποιούνται αναπερίπτωση. Αυτό είναι ε, ένα οικονομικό πλεονέκτημα βέβαια. Ε, και ήμασταν σε θέση ε, να πούμε ότι με ικανοποίηση έχουμε πληρώσει το, το, το έργο μας. Τώρα στο μέλλον δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Σε περίπτωση που αλλάζουν πολλοί αποστολές και αλλάζουν και ε, υπάρχει μια ε, σύνδεση στρατιωτικού και πολιτικού σκέλους. Θα πρέπει να διατηρηθούν οι γνώσεις οι τα διδάγματα που έχουν εξαχθεί και ε, να δρούμε και σε αποστολές ε, άμεσης, επίγουσες, όπως σε περίπτωση θεομηνιών. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε το θέμα αυτό ρεαλιστικά, ε, νυφάλαια, με ένα σαφή ορισμό, το τι επιθυμούμε από πλευράς λειτουργίας πλέον και όχι δομών. Πώς να λειτουργούμε και στη συνέχεια να αξιολογήσουμε αν αρκεί να βελτιώσουμε του υφισταμένους μηχανισμού ή μήπω χρειάζονται πιο φιλόδοξε λύσει. σε ό,τι αφορά την αγορά της ε, άμυνας και την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα εξακολουθεί να προωθεί την διαφάνεια και το ευρύτερο άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς χάρη στους κώδικες συμπεριφοράς για τις προμήθειες στην άμυνα, τον ε, κώδικα καλών πρακτικών για την ε, φοδιασμό και σε ό,τι αφορά τον κώδικα για τις προμήθειες, αμυντικές προμήθειες, από όταν άρχισε να εφαρμόζεται το 2006 πάνω από 1.600 ε, συμφωνίες προμηθειών των οποίων εξή ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ε, ανατέθηκαν και η συνολική τους αξία ήταν πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ και οι διασυνοριακές προμήθειες από το 20% το 2007 φτάσαν στο 47% το 2010 εξ όσων αυτά είναι τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Ο οργανισμό συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει και να καταστήσει διαφανή και ανταγωνιστική την αγορά στρατιωτικών εξοπλισμών με βάση την οδηγία για την υπογραφή κάποιων συμβάσεων προμηθειών στον τομέα τη άμυνα και τη ασφάλεια που θα ενσωματώσουν στην εθνική του νομοθεσία τα κράτη-μέλη μέχρι το καλοκαίρι του 2011. Και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, η βιομηχανική και τεχνολογική βάση για την, άμυνα, την ευρωπαϊκή άμυνα αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των στρατιωτικών ε, ικανοτήτων της Ευρώπης, ειδικότερα για τον τομέα της τεχνολογίας, για την οποία δεν θέλει να εξαρτάται από εξωτερικές προμήθειες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα, βεβαίως το, η όλη δομή θα, θα επηρεαστεί από τις περικοπές των αμυντικών δαπανών. Γι' αυτό θα χρειαστεί να μειωθούν οι επικαλύψεις στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη και να υπάρξει μεγαλύτερος εξορθολογισμός. Οι εθνικές βιομηχανίες δεν μπορούν να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους αν μειωθούν οι εθνικές παραγγελίες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και στον τομέα των κρατικών προμηθειών. Θα χρειαστεί λοιπόν να εξασφαλιστεί μια μετάβαση προοδευτική σε μια τεχνολογική και βάση για, μια, ε, για την ευρωπαϊκή άμυνα τα αεροπορικά συστήματα θα είναι το πρώτο πιλωτικό σχέδιο. Οι εργασίες του οργανισμού για, την, για την, ίσους ανταγωνιστικούς όρους θα συμβάλλει στην ε, διαφάνεια και στο άνοιγμα ε, των αγορών και υπάρχουν ε, σαφείς προϋποθέσεις ε, για την πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά, έλεγχος των ξένων επενδύσεων από το κράτος και ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ορισμένοι από εσά αναφερθήκατε στις ερωτήσεις σας στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και πολύ δικαίως επιμείνατε σε αυτή τη σχέση που είναι σημαντική και η οποία καθίσατε όλο και πιο σημαντική προκειμένου να αποφευθούν ε, συνέπειες ε, στην ανάπτυξη των ε, ικανοτήτων και από δημοσιονομική άποψη αλλά και για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στους δύο οργανισμούς. Θυμίζω ότι η αποστολή που ανατέθηκε στην κυρία Άστον γιατί έχει σκοπό να εξασφαλίσει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των κρίσεων. Και πέρα από αυτό δεν πρέπει, πρέπει να αναπτύξουμε και μια ουσιαστική πολιτική σχέση ανάμεσα στους δύο οργανισμούς. Ορισμένοι από εσά ο κύριος Νταφ και ο κύριος Τάνοκ ειδικότερα αναφέρθηκαν στο θέμα ε, στο Κυπριακό στις σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας που οπωσδήποτε είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η κυρία Άστον έχει αναλάβει σχετικές δεσμεύσεις, αλλά αναμένοντα την επίλυση, οι δύο πλευρές πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη ευελιξία για να δημιουργηθεί μια επικοδομητική δυναμική. Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση, Ορισμένοι από εσά αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα. Το στοιχείο, είναι στοιχείο κλειδί για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης στο σύνολό τη και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ε, πρόθεση της ΕΠΑ. Το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Άμυνας, κατά την άποψή μας, παίζει σημαντικό ρόλο. Η, σχολή, ε, Ευρωπαϊκή Σχολή Άμυνας είναι πολύ σημαντική για στον τομέα της κατάκτησης. Ορισμένα αναφέρθηκαν και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας για τη διαχείριση των κρίσεων και πάλι. Σας θυμίζω τη συνεργασία με τη Ρωσία στην, στο Τσάτ και στην Κεντρική Αφρική με τη Γιορφόρ και ας μην ξεχνάμε τον διάλογο που συνεχίζεται στα πλαίσια τη της Κέρκυρας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και, του, και Ρωσίας πρέπει οπωσδήποτε να διευρυνθεί και να ενισχυθεί. Τώρα, Υπήρξαν και, αναφέρθηκαν ε, και ορισμένοι ομιλητέ του Αφγανιστάν. Τα κράτη μαέλη αυξάνουν τη συνεισφορά του ε, στην αποστολή, στην επιχείρηση στο Αφγανιστάν που αντιμετώπισε δυσκολίε στην αρχή αλλά τώρα πλέον και έχει καταστεί πιο αποτελεσματική σε συνεργασία με την αποστολή του ΝΑΤΟ για την κατάρτιση των ε, δυνάμεων ασφαλεία. Οι δύο αποστολέ αυτέ αλληλοσυμπληρώνονται και πολύ σωστά είπατε ορισμένοι από εσά σήμερα πολύ σωστά είπατε ότι αυτή είναι μια προτερότητα και υπάρχει και μια άλλη προτεραιότητα που συνδέεται με αυτή, η, κατάρτιση των δυνάμεων ασφαλείας του Αφγανιστάν, ώστε να αναλάβουν οι ίδιοι πλέον τις ευθύνες τους. Κύριε, Πρόεδρε, αυτά ήταν κάποια στοιχεία απάντησης που θέλησα να συνεισφέρω στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ να το χειροκροτήσουμε τον κύριο Σαστέλ όπως το αρμόζει ε, και στο έργο του και στις εξαντλητικές και πλήρες απαντήσεις που μας έδωσε. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και σημαντικό το θέμα της ενίσχυσης της ε, ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό σήμερα είχαμε μια πρώτη συνάντηση, αλλά η συνεργασία μας με βέβαιο θα συνεχιστεί και με τρόπο πιο εντατικό και πλήρη τους επόμενους μήνες και έτσι. Το επόμενο μέρος τώρα στη συνεδρίασή μας προβλέπει την εδραίωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και η ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου τώρα είναι ένα θέμα το οποίο θα προεδρεύσει ο ε, κύριος Νονζόν, πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Εγγύηση λοιπόν της νομιμότητας με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της ΕΠΑ. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε στο δεύτερο τμήμα αυτής της συνεδρίασης για την νομιμότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου της ε, ΕΠΑ ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο των ε, κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων μας εδώ, στο Στρασβούργο και στις ε, πρωτεύουσές μας. Το θέμα της, παρακολούθησης, της κοινοβουλευτικής παρακολούθησης της ΕΠΑ είναι ιδιαίτερα επίκαιρο λόγω δύο γεγονότων. Αφενός, την καταγγελία της σύμβασης, τη ε, λύση, τη λύση της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης και την έναρξη ισχύω του, της συνθήκης της τη της οποίας το πρωτόκολλο 1 καλεί της, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να καθορίσουν από κοινού την προώθηση μιας διακοινοβουλευτικής συνεργασίας που θα είναι τακτική και αποτελεσματική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από αυτές τις ε, συνταγματικές επιταγές υπάρχει και μια πολιτική διάσταση που είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ΕΠΑ, να το θυμίσουμε αυτό, δεν είναι απλά μια φιλοδοξία που αναφέρεται σε μια συνθήκη, αλλά μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία σήμερα τη στιγμή που μιλάμε εκφράζεται μέσα από 14 πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές που έχουν αναπτυχθεί σε ζώνες κρίσης ανά τον κόσμο και υποστηρίζεται εδώ στις Βρυξέλλες και στις πρωτεύουσές μας από εκατοντάδες άτομα που που αποτελούν στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Χρειάζεται λοιπόν μια αυξανόμενη παρακολούθηση και προσοχή ε, για τις εξελίξεις αυτές εκ μέρους των ε, ε, κοινοβουλίων για τα άτομα, τους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε αυτές τις επιστολές και το κοινό, διότι οι συμπολίτε μας γνωρίζουν πολύ λίγα πράγματα για αυτές τις αποστολές, για αυτές τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο όνομά τους. Και όταν κάτι και όταν ενημερώνονται για αυτές τις υποστηρίζουν ένθερμα. Πρέπει λοιπόν ως κοινοβούλια να εξασφαλίσουμε την επαφή ανάμεσα στους υπαλλήλους και, ε, που συμμετέχουν σε αυτές τις αποστολές και τους πολίτες για τους οποίους διεξάγονται αυτές οι αποστολές. Η ε, συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να καλύψει ορισμένα, ορισμένα σημεία στα οποία θα αναφερθώ και εγώ, αλλά και πολύ πιο λεπτομερώς ο συνάδελφο Μπροκ, αλλά σαν μια εισαγωγή θα ήθελα να θυμίσω ότι όλοι γνωρίζουμε το ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα της τομέα της άμυνας και τα προβλήματα κυριαρχίας ε, που προκύπτουν. Τούτου λεχθέντος θέλω να επιμείνω στο γεγονός ότι η ΕΠΑ διεξάγει πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις. 14 που ανέφερα που βρίσκονται υπό εξέλιξη, 12 είναι πολιτικές επιχειρήσεις. 23 που έχουν ξεκινήσει από το 99 σε αυτές τις 23 λοιπόν αποστολές, 15 ήταν πολιτικού χαρακτήρα, 7 στρατιωτικές αποστολές και μόνο μία ήταν η κοινή πολιτικο-στρατιωτική αποστολή. Μιλάμε λοιπόν ότι, οι πολιτικές αποστολές είναι, αποτελούν την πλειοψηφία των αποστολών που ε, διεξάγονται στα πλαίσια της ΕΠΑ, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό ε, είναι απαραίτητο να συμμετέχει στη διαδικασία της απόφασης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τακτική διαβούλευση βάσει του άρθρου 36 ε, γίνεται μεταξύ της ΥΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάντοτε για τα θέματα της ΕΠΑ. Προσθέτω επίσης ο κύριος Αλμπερτίνη και ο συνάδελφος Λαμασούρ και εγώ ο ίδιος πέντε φορές το χρόνο συνεδριάζουμε ε, ε, με το Συμβούλιο, με το Συμβούλιο για όλες τις, ε, τις επιχειρήσεις και τις αποστολές που βρίσκονται, που βρίσκονται υπό εξέλιξη, τις οποίες και αναλύουμε και εξετάζουμε σε όλες τις λεπτομέρειες. Μιλάμε λοιπόν για μια πολύ στενή και επικοδομητική συνεργασία. Αυτά ήθελα να πω ε, σαν σύντομη εισαγωγή στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Οντρέ Φλαό θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Ντονίμ Κάρν που είναι μέλος Συμβουλευτικής ε, ε, Επιτροπής για τα ευρωπαϊκά ζητήματα που θα λάβει το λόγο αμέσως μετά τον συνάδελφο Ελμάρ Μπροκ που είναι ο εισηγητής για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκών και ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Ελμάρ, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ ε, για την εισαγωγή. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας και τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάτης εκπροσώπου που είναι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε πλέον μια νέα κατάσταση στο θέμα της νομιμότητας των πολιτικών αποφάσεων σε επίπεδο εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν συνέπεια της συνθήκη διότι με τη δημιουργία της θέσης της υπάτης εκπροσώπου οι κοινοτικές ε, σχέσεις που είναι μερίδα του λέοντος πολιτικής ε, γειτονίας, ε, εξωτερικές βοήθειες, αναπτυξιακή βοήθεια και εξωτερικό εμπόριο παρακαλώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο κοινοτικών αρμοδιοτήτων ως προς τις εξωτερικές σχέσεις. Και η ΚΕΠΑ και η ΕΠΑ είναι οργανωμένοι διακυβερνητικά. Η ύπατη εκπρόσωπος δραστηριοποιείται και στα δύο όργανα. Προεδρεύει στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, αλλά και αντιπρόεδρο ταυτόχρονα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση εργάζεται και για τι δύο αυτέ υπηρεσίε, αλλά δεν έχει ε, δυνατότητα λήψη αποφάσεων. Τι αποφάσει τι παίρνει είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε το Συμβούλιο. Παραμένει. Δηλαδή, η υπηρεσία αυτή έχει στόχο να πλαισιώνει την ύπατη εκπρόσωπο και να την ε, καθιστά ε, ικανή να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά της και να δημιουργούνται και συνέργειες από την συνεργασία εκεί των υπηρεσιών ε, έτσι ώστε να έχουμε σωστή πολιτική στο μέλλον. Τώρα είπατε εκπρόσωπος ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως Πώς να... Κάποιος έχει αφήσει το ξυπνητήρι του Blackberry ανοιχτό, αλλά έχω ξυπνήσει. Πείτε του σας παρακαλώ. Λοιπόν, τι έλεγα. Η ύπατη εκπρόσωπο λοιπόν είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως κάθε άλλος επίτροπος υπόκειται σε ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, και σε έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να γίνει μέλος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό τι σημαίνει. Λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Accountable to European Parliament το λένε αυτό στα αγγλικά. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να την καθαρέσει, όπως και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό και μόνο, ε, κατά κάποιο τρόπο, αλλάζει και τη σχέση που έχει η κυρία Άστον με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα αυτό. Άλλο θέμα τώρα. Ο πολιτικός έλεγχος. Δεν είναι στο παλιό πλέον άρθρο 21, αλλά στο μέλλον η σύνολη υπηρεσία υπόκειται στον πολιτικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είπα ότι εκπρόσωπος είναι υποχρεωμένη να αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τη συνθήκη και από τα όσα δήλωσε το Κοινοβούλιο για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Δράσης. Και αν κολλείεται η ίδια να αναφέρει στην Ολομέλεια τη αρμόδια επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να την αντικαθιστούν επίτροποι και πάλι και με τη μεικτή ιδιότητα όταν μιλάμε για το Αφγανιστάν ας πούμε που έχει να κάνει με την κανονική κοινωνική, κοινοτική βοήθεια συγγνώμη, ε, και το στρατιωτικό και το πολιτικό θα πρέπει να είναι επίτροποι επαναλαμβάνω που είναι υπόλογοι 100% στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε περιπτώσεις τώρα αμυγής της ΚΕΠΑ μπορούν να την εκπροσωπούν μόνο ε, οι εκπρόσωποι του τρίου στο, Υπουργό, ε, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Δηλαδή, υπουργοί, ε, μία από τις τρεις προεδρίες. Στο μέλλον, λοιπόν, δεν συζητούν μόνο, είπατε εκπρόσωπος και το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μόνο είπατε εκπρόσωπος ή κάποιο που την αντικαθιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν και να αναφέρουν για τις κινήσεις τους. Επί της ουσίας τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι απλώς γενική διαβούλευση και ενημέρωση, αλλά πριν από σημαντικές αποφάσεις για στρατηγικές και για αποστολές, το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή Εξωτερικών θα πρέπει να λέει τη γνώμη της. Και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων είμαστε ε, εμείς εξειδικευμένοι στις, στην Επιτροπή Ασφάλειας Και το Κοινοβούλιο ε, έχει και πενταμελή επιτροπή, όπου προεδρεύει ο πρόεδρος της ε, ε, Επιτροπής Εξωτερικών, που έχουν και τη δυνατότητα να διαβάζουν και να κοιτούν τα έγγραφα και να ενημερώνουν και την κυρία Άστον. Δηλαδή, είναι δεδομένος ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, όπως συμβαίνει και στα εθνικά κοινοβούλια. Πέρα λοιπόν από το δεδομένο πολιτικό έλεγχο και στο συμπαγή στο μέλλον, οι πρέσβει τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποχρεούνται να λογοδοτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούν να προσκαλούνται ανα πάσα στιγμή και να υπόκεινται σε ένα είδο ακρόαση ανταλλαγή απόψεων πριν αναλάβουν τα καθήκοντά του, τα διαπιστευτήρια. Δεν θα το κάνουμε βέβαια για τον καθένα, αλλά το δικαίωμα το έχουμε και το έχουμε ήδη πράξει σε μερικέ περιπτώσει. Δηλαδή, και πάλι εδώ ε, έχουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και ανεξαρτήτως των καθηκόντων του καθενός. Άλλο θέμα τώρα. Θα πρέπει να πούμε ότι το σύνολο κεφάλαιο του προϋπολογισμού μπαίνει τώρα στη συναπόφαση του Κοινοβουλίου. Άρα και ο προϋπολογισμός για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Και ταυτόχρονα έχουμε λοιπόν και τον δημοσιονομικό έλεγχο από το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ο συνολικός ε, διοικητικός, λειτουργικός προϋπολογισμός και ο ε, εξωτερικός προϋπολογισμός ελέγχονται από το Κοινοβούλιο. Τα διαχειρίζεται αυτά οικονομικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα και εδώ είναι πλήρης ο έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα οικονομικά. Δηλαδή, παντού όπου είναι ευρωπαϊκέ κοινοτικέ οι αρμοδιότητε, στην ουσία εμεί έχουμε καλύψει αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα και δεν υπάρχει το κενό. Τώρα όμω συμβαίνει και το εξή Στα στρατιωτικά, που και αυτά είναι συστατικά τη εξωτερική ε, δράση υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορισμένες αποφάσεις είναι μετατοπισμένες, είναι στα χέρια των Εθνικών Κοινοβουλίων τα Εθνικά Κοινοβούλια έχει τη δυνατότητα βέβαια να ελέγχει σε όλους τους τομείς τις κυβερνήσεις της κάθε χώρας. Τις κυβερνήσεις ως μέλη του Συμβουλίου. Αυτό είναι δεδομένο έτσι κι αλλιώς. Ελέγχει το Κοινοβούλιο. Πλην όμως θα πρέπει τα Κοινοβούλια να το πράττουν κιόλα. Κάτι άλλο που ισχύει για τη δική μου χώρα, όταν στέλνουμε ένοπλες δυνάμεις, υπάρχει επιφύλαξη του Κοινοβουλίου. Πρέπει να δώσει την έγκρισή του το Κοινοβούλιο. Και εγώ διαφωνώ να καταργηθεί αυτό. Διότι δεν μπορούμε να στέλνουμε ένοπλες δυνάμεις εκτός κοινοβουλευτικού ελέγχου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν το έχει αυτό το δικαίωμα. Μόνο τα εθνικά κοινοβούλια, ανάλογα με τα συντάγματα της κάθε χώρας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε ευρωστρατό αμέσως. Γιατί με τον ευρωστρατό κανονικά θα συνδεόταν αυτή η εξουσία, ότι η εντολή η αλυσίδα της διοίκησης θα πρέπει να έχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα και αυτό είναι ε, κάτι που δεν είναι του παρόντος. Δεν μπορεί ας πούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει ότι ο στρατός μιας χώρας θα πρέπει να πάει κάπου και να διαφωνεί το Κοινοβούλιο της ίδιας της χώρας και να ληφθεί η απόφαση παρά τη βούληση της κυβέρνησης ή της βουλής της χώρας. Αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, και ένα τελευταίο είναι ε, η χρηματοδότηση των εθνικών ενόπλων δυνάμεων που συμμετέχουν σε αποστολές. Είναι και αυτό θέμα εθνικών κοινοβουλίων και ο κοινοβουλευτικό έλεγχο αναλογεί σε αυτά τα κοινοβούλια. Λοιπόν, είναι σαφής ο διαγωνισμός. Ό,τι έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό επίπεδο, με το κοινοτικό επίπεδο, είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενώ μια σειρά θεμάτων είναι σαφώς ε, στην εξουσία των Εθνικών Κοινοβουλίων και στον έλεγχο του προπολογισμού. Δεν υπάρχει κανένα κενό εδώ νομικό που να χρειάζεται να καλυφθεί. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί νέα συνέλευση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τα άλλα δεν θα ήταν πρόθυμο και ουσιαστικά δεν θα ήταν και νομικά σε θέση να ε, ε, μεταθέσει αρμοδιότητες σε μια τέτοια συνέλευση που δεν προβλέπεται από καμία συνθήκη. Και υποθέτω και τα εθνικά κοινοβούλια δεν θα ήταν πρόθυμα να το πράξουν σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμεί. Καλύτερο συντονισμό και καλύτερη ενημέρωση να έχουμε. Αυτό δεν γίνεται με μια συνέλευση που θα συσταθεί και θα συνεδριάζει άπαξ ετησίω με μεγαλόστομε ομιλίε και δηλώσει. Με μια γραμματεία που θα έχει και τη φιλοδοξία να πτύξει να κάνει δικέ τη εκθέσει, που έτσι κι αλλιώ δεν θα τι διαβάζει κανένα γιατί δυσκολευόμαστε να διαβάζουμε και τι δικέ μα. Και θα δημιουργήσουμε εκεί πέρα ένα πομπόδες κατασκεύασμα που δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα για λήψη αποφάσεων από καμία συνθήκη. Γιατί αυτά παραμένουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια, το καθένα ξεχωριστά. Και δεν μπορούν τα Εθνικά Κοινοβούλια να μοιραστούν μεταξύ τους τις δικές τους αρμοδιότητες. Κάθε κοινοβούλιο έχει δεδομένες αρμοδιότητες και εξουσίες. Λοιπόν, εάν θέλουμε να λάβουμε σοβαρά ε, υπόψη το ρόλο μας και να τον ασκήσουμε απέναντι στην ύπατη εκπρόσωπο στα ε, Συμβούλιο και το ίδιο να ισχύει για τα Εθνικά Κοινοβούλια απέναντι στις εθνικές κυβερνήσεις συνιστάται να έχουμε ανταλλαγή απόψεων, ανταλλαγή ενημέρωσης για να μην μας χρησιμοποιεί κανένας για να μας μεταχειριστεί ε, τον ένα βάρος του άλλου. Εδώ έχουμε συναντήσεις, αλλά δεν θα πρέπει να έρχονται κάποιοι, γενικώ κάποια μέλη, αλλά εκείνοι που παίρνουν τι αποφάσει στι επιτροπέ εξωτερικών και στι επιτροπέ αμήνη. Όχι κάποια μέλη, οι πρόεδροι, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ε, συγκεκριμένοι φορεί των κοινοβουλίων και συγκεκριμένα πρόσωπα. Και αυτό γίνεται μόνο σε συνεργασία με τι επιτροπέ εξωτερικών του εκάστοτε κοινοβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε και νέα γραμματεία, μπορεί να το κάνει η γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί σε κάθε γραμματεία, κάθε ε, Επιτροπής Εξωτερικών κάθε Εθνικού Κοινοβουλίου έχουμε ένα πρόσωπο που είναι ε, ο συνομιλητής μας, ο σύνδεσμός μας και προφορικά και γραπτά μπορούμε να συνεννοούμαστε και να επικοινωνούμε και όπως είπε και, κύριος, και το έκανε ο κύριος Αλμπερτίνη και εγώ στο παρελθόν που είχα διατελέσει πρόεδρος Είχαμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ανταλλαγέ απόψεων και στι Βρυξέλλε και φρονώ ότι πρέπει να οργανωθεί αυτό και να συστηματικοποιηθεί και να ενταθεί. Όχι να βγαίνουμε και να βγάζει ο καθένα ένα λόγο, τι ωραία που είμαστε πάλι μαζί όλοι εδώ συγκεντρωμένοι. Α πούμε, τι θα γίνει με τον αμυντικό οργανισμό. Defense Agency είναι υπό τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά εκεί υπάρχουν θέματα προμηθειών και άλλα που παραμένουν εθνικές αρμοδιότητες για τις αμυντικές δαπάνες. Και αν θέλουμε να έχουμε ενιαία πολιτική για την αμυντική βιομηχανία και για τις προμήθειες στην άμυνα, καλό θα είναι να ενημερώνομαστε, να συνεννοούμαστε για να μην γίνονται διάφορες κινήσεις. Ούτε μεγάλες εκδηλώσεις μια φορά το χρόνο να έρχεται η κυρία Άστον επαιτειακά να βγάζει μια ομιλία και μετά να λέει «Μα τι θέλετε, ωραία σας ενημέρωσα και πάει, αυτό διεκπεραιώθηκε αφού ήρθα». Όχι. Δεν θα πρέπει να την αφήσουμε να πάρει αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου δεν πιέζει και ο χρόνος. Ακόμα δεν έχει οριστεί τίποτα. Ελπίζουμε να φροντίσει να έρθει την 1η Δεκεμβρίου η κυρία Άστον. Ε, σε επίπεδο όμως ε, τεχνικό να έχουμε καλύτερη συνεργασία για να ανταποκριθούμε καλύτερα στο ρόλο μας και στα καθήκοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μπροκ. Ο κύριος Ντουκάρμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και με τη δική μου σειρά θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του κυρίου Πλαού που είναι, ε, προέρχεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του ε, Βελγίου και εκπροσωπεί το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ε, επί Ευρωπαϊκών Θεμάτων, της Συμβουλευτικής Επιτροπής επί Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Θα ήθελα με τη σειρά μου να μιλήσω για τις νέες προκλήσεις της, στην ΕΠΑ μετά τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον ε, κύριο Αλμπερτίνη, πρόεδρο της ΑΦΕΤ και εσάς ε, κύριε Ντανζόν, που είσαστε πρόεδρο της Υποεπιτροπή Άμυνα και Ασφάλειας που, λάβατε αυτή, που αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα το οποίο χρήζει βάθυνσης τόσο από τα, Ευρωπαϊκά κοινοβούλια, Εθνικά Κοινοβούλια όσο και από το Ευρωπαϊκό σε σχέση με την πολιτική, το πολιτικό σκέλος της μεταρρύθμισης αυτής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Έλμαρ Μπροκ για τα επικοδομητικά του σχόλια διότι μας μίλησε για την συλλογιστική που μας απασχολεί και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να υπάρχει μία εγγύηση της νομιμότητας μετά από κοινοβουλευτικό έλεγχο της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και ως προς τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος αυτής της ευρωπαϊκής δύναμης και αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των Εθνικών. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που προσδίδουμε ως Βελγικό Κοινοβούλιο στο όλο θέμα. Ε, ασκούμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως γνωρίζετε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων που είναι ε, παρόντες εξ ονόματος του Βασιλείου του Βελγίου. Στην ΚΟΦΑΚ η ΚΟΦΑΚ μάλλον, που είναι η διάσκεψη για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, θα ε, λάβει χώρα στο Βέλγιο στις 18 και 19 Οκτωβρίου και η ύπατη εκπρόσωπος θα εκφράσει τις απόψεις της. Θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας από τα κράτη-μέλη και στις 25 και 26 Οκτωβρίου στο Παλέ θα διοργανωθεί η 44η ε, Σύνοδος της Κόζακ και πιστεύω ότι η ΕΠΑ και η ΚΕΠΑ θα μας απασχολήσουν στα πλαίσια της 44ης διάσκεψης της ΚΟΖΑΚ και θα πρέπει όλοι να απαντήσετε σε ένα ερωτηματολόγιο. Με βάση τις απαντήσεις η γραμματεία της ΚΟΖΑΚ θα προβεί σε ένα συγκεφαλαιωτικό έγγραφο και θα δημοσιευτεί στα πλαίσια της ΚΟΖΑΚ. Άρα οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων στη, το 2010 θα μας μιλήσουν για τον ρόλο της ΕΠΑ και των Εθνικών Κοινοβουλίων και γι' αυτό ως Προεδρία θεωρούμε ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να ελέγχουν μελλοντικά την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας καθώς και την εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό η διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε εντολή στο Βελγικό Κοινοβούλιο μαζί με το Ευρωπαϊκό να συντάξουν μία πρόταση σε σχέση με την νομιμότητα και τον έλεγχο αυτό που θα υποβληθεί στην επόμενη διάσκεψη των Προέδρων που θα ε, γίνει το 2011 την Άνοιξη. Επίσης, μετά από τη σύνοδο στη Μαδρίτη, η Κόζακ, μετά τη λήξη των εργασιών της, τόνισε ότι λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιάζοντα χαρακτήρα αυτών των εργασιών, η Κόζακ υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων για, την, για τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής και κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Άρα υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος, θα υπάρξει κοινοβουλευτικός έλεγχος μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Και αυτό αποτελεί ένα νέο στάδιο για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Γι' αυτό στις 31 Μαρτίου 2010 αποφασίσαμε να καταγγείλουμε την ε, παλαιότερη συνθήκη και μέσα στα πλαίσια της ρήτρα αμοιβαία συνδρομής στο άρθρο 41.7 της Συνθήκης της Λισαβόνας θεωρούν τα κράτη-μέλη ότι αρχίζει μία νέα φάση για την ΕΠΑ θέτοντας τέλος στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση που είχε συσταθεί το 1954 και έτσι η κοινοβουλευτική συνέλευση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα δρά πλέον και θα ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό. Τον Ιούνιο του 2011 λοιπόν λήγουν οι εργασίες της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα παραμένει ανοιχτό το θέμα του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού ελέγχου στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας. Πώς ε, θα ε, επανδρωθεί αυτό το πλαίσιο και πώς θα λειτουργήσει. Άρα τα εθνικά κοινοβούλια των 27 κρατών μελών θα πρέπει να συζητήσουν επιθεμάτων ΕΠΑ και να ορίσουν την ε, λειτουργία ελέγχου και εποπτείας. Πώς θα λειτουργήσουν μελλοντικά οι ΚΕΠΑ και ΕΠΑ. Στο briefing αυτό ορίστηκε ότι η ΑΦΕΤ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ε, διοργανώνει μία σύνοδο με τα Εθνικά Κοινοβούλια για τη λειτουργία της ΕΠΑ και της ΚΕΠΑ. Άρα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτό το διτό δημοκρατικό έλλειμμα. Θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε τη διακριτική ευχαίρεια λήψη αποφάσεων μέσα στα πλαίσια της ΕΠΑ και επίσης τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να ανταποκριθούν στη λήψη αποφάσεων ως προς τη λειτουργία της ΕΠΑ και της ΚΕΠΑ. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε και να επαυξήσουμε τη νομιμότητα των αποφάσεων μέσα στα πλαίσια ΕΠΑ και ΚΕΠΑ. Πώς να μην έχουμε έναν μεγάλο κατακαιρματισμό της εποπτείας και του ελέγχου των δύο αυτών πυλώνων της ΕΠΑ και της ΚΕΠΑ και να υπάρχει μεγάλη ορατότητα και συνέχεια καθώς και συνοχή. Πώς μπορούμε να συνδράμουμε έτσι ώστε να υπάρχει αποδοτικότητα με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αυτό, αυτά τα θέματα μας απασχολούν επί της ουσίας και υπάρχουν, υπάρχει ένας ε, εμπειρογνώμενος ο οποίος θα αποφανθεί επί του θέματος, ο κύριος Αντρέ Τζιμουλέν από το Βελγικό Κοινοβούλιο, από τη Βελγική Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο πρόεδρος Ντάνζον αναφέρθηκε στη συνθήκη της Λισαβόνας η οποία αποτελεί ε, τον μύτο που θα μας οδηγήσει στο άρθρο 36 όπου γίνεται διαβούλευση με την ύπατη εκπρόσωπο για τις βασικές επιλογές επί ΕΠΑ και ΚΕΠΑ, για να δούμε πώς ενισχύονται και εξελίσσονται αυτές οι πολιτικές. Η ύπατη εκπρόσωπος λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών. Και δύο φορές το χρόνο γίνεται μία συζήτηση για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί ως προς την κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Αν λάβουμε υπόψη το άρθρο 9 του πρωτοκόλου, όπως είπε και ο κύριος Μπροκ ως προς το ρόλο των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, βλέπουμε ότι αναγράφεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια ορίζουν από κοινού έναν διακοινοβουλευτικό διάλογο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δυνάμει του άρθρου 10, μία διάσκεψη διοργανώνεται η οποία έχει ε, διακοινοβουλευτικό χαρακτήρα για να συζητηθούν θέματα εξωτερικής πολιτικής και κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει ανάγκη συνέχειας έτσι ώστε η ΕΠΑ και η ΚΕΠΑ να υφίστανται έναν δύο κοινοβουλευτικό διάλογο από τα 27 κράτη-μέλη, κάτι το οποίο αναγνωρίζουν πλέον και τα εθνικά κοινοβούλια. Θα ήταν λυπηρό να μην τεθεί κάτι τέτοιο σε εφαρμογή δυνάμει της συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να μην παλινοδίσουμε ως προς τον ρόλο μας στον τομέα της ενίσχυσης της άμυνας και ασφάλειας, έτσι ώστε να δώσουμε τη σκητάλη και στην κοινή γνώμη. Τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι αρμόδια για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό, εκεί όπου προβλέπεται. Υπάρχουν όμως και στοιχεία τα οποία δεν έχουν καθοριστεί επακριβώς. Μιλάμε για αύξηση των προνομίων ελέγχου της νομιμότητας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα διαγράφονται διάφορες ε, εναλλακτικά σενάρια ελέγχου ΕΠΑ και ΚΕΠΑ. Ήδη πολλά εθνικά κοινοβούλια εκφράστηκαν επί του θέματος είτε σε επίπεδο Επιτροπής ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων είτε σε επίπεδο Ολομελίας. Βεβαίως κάθε πρόταση είναι διαφορετική ως προς τη σύνθεση των αντιπροσωπιών, την χρηματοδότηση, την περιοδικότητα των συνεδριάσεων και ούτω καθεξής. Δεν μπορώ να αναφερθώ πιο διεξοδικά στις ε, θέσεις που έχουν εκφράσει όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να συνδράμουμε σε αυτή τη συζήτηση τονίζοντας ορισμένους σημαντικούς άξονες με βάση την ε, κοινοβουλευτική συνέλευση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους έγινε ε, λόγος για συνεχή έλεγχο της ΕΠΑ και ΚΕΠΑ δυνάμει της συνθήκη, του πρωτοκόλου 1 της συνθήκης της Λισαβόνας που έχει κυρωθεί από τα 27 κράτη-μέλη ε, και από το Ευρωπαϊκό. Και οι εθνικές αντιπροσωπείες θα εκπροσωπούνται ε, αναλογικά και, στην, ε, ε, και στα πλαίσια της ΕΠΑ. Θα υπάρχει λοιπόν συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται ο ρόλος των κρατών μελών στον προσδιορισμό της ΕΠΑ και της ΚΕΠΑ. Αυτή η μόνιμη διάσκεψη θα συντάξει μια ετήσια έκθεση και θα απαρτίζεται από δύο επιτροπές, τη μία για τις εξωτερικές υποθέσεις και τη δεύτερη για θέματα άμυνας και ασφάλειας. Και έτσι θα ασχοληθούμε και με θέματα εξοπλισμού. Επίσης θα ε, συνδράμεται από μία ε, γραμματεία, η μία θα είναι μόνιμη και η άλλη περιοδική και θα χρηματοδοτείται από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Άρα θα συνεργαστεί με την COPS και θα προβλέπονται δύο συνεδριάσεις ανά στις ε, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Επίσης, θα υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση και ε, επιμελητιακή βοήθεια και θα καλύπτεται και το κόστος των μεταφράσεων. Επίσης, θα υπάρχει και μια διεύθυνση ευρωπαϊκών ε, σχέσεων η οποία θα συνδράμει στο όλο έργο. Μία, ένας δεύτερος άξονας αφορά την ανάληψη της ΕΠΑ και της ΚΕΠΑ από την ΚΟΖΑΚ. Θα προβλέπονται έκτακτες συνεδριάσεις σε αυτή την περίπτωση και ίσως αλλάξει και ο εσωτερικός κανονισμός. Αυτή είναι η δεύτερη εναλλακτική που θα μπορούσαμε να προβάλλουμε. Ίσως και άλλοι ε, συμμερίζεστε αυτή τη μινιμαλιστική προσέγγιση. Μία τρίτη εναλλακτική αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της ΕΠΑ και ΚΕΠΑ στο φόρουμ συνεργασίας, στα φόρα συνεργασίας που υπάρχουν, δηλαδή ε, τις ε, ε, Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων ή από την Κόντακ. Σε αυτή την περίπτωση τα φόρα αυτά θα αποφασίσουν για την μορφή ελέγχου της νομιμότητας των ΕΠΑ και ΚΕΠΑ. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος θα μπορέσει να λάβει χώρα είτε στα πλαίσια της ΚΟΦΑΚ ή της ΚΟΝΤΑΚ η οποία θα επεκταθεί, θα διευρυνθεί. Θα έχουμε έξι βουλευτές ανακράτος μέλος και έξι μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και την συνδρομή μιας γραμματείας θα υπάρχει μια περιοδικότητα και θα γίνεται μια συνεδρίαση ανά Το παράδειγμα που σας έφερα σχετίζεται με μια πρόταση ψηφίσματος της Γαλλικής Γερουσίας. Υπάρχουν και άλλα κοινοβούλια που μίλησαν για μια νέα διάρθρωση η οποία ε, θα αφορά όχι μόνο την ε, συνδρομή της αλλά και της ΚΟΝΤΑΚ. Αυτή η πρόταση απορρέει από τις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων, ε, ιδιαίτερα αυτήν του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης υπάρχει και η τρίτη εναλλακτική που προέβαλε η Ιταλική Γερουσία για τον έλεγχο της ΚΕΠΑ ΚΕΠΑ όπου ε, συνδράμουν και τα, ε, ευρωπαϊκά, και τα, ευρωπαϊκά, ε, τα εθνικά κοινοβούλια και το ευρωπαϊκό. Και βεβαίως εκεί που υπάρχει Βουλή Αντιπροσώπων και Γερουσία θα συμμετέχουν και τα δύο σώματα. Οι συνεδριάσεις αυτές θα γίνονται στις Βρυξέλλες κάθε εξάμηνο, μία φορά το εξάμεινο και βλέπετε λοιπόν ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη συλλογιστική είδη και υπάρχει πληθώρα προτάσεων. Έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε όλες αυτές τις ε, δομές επαρκώς. Αλλά υπάρχουν και ε, διάφορες εναλλακτικές μέσα ε, στα πλαίσια του κάθε άξονα προτάσεων η Επιτροπή Άμυνας θα ήταν μια, ε, άμυνας και ασφάλειας θα είναι μια επιτροπή και όχι υποεπιτροπή πλέον. Και βεβαίω οι θέσεις διαφέρουν από ένα κοινοβούλιο στο άλλο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ενισχυθεί ο έλεγχος της νομιμότητας των ΕΠΑ και ΚΕΠΑ γίνονται συζητήσεις αλλά δεν έχουν αποκρισταλωθεί προτάσεις. Στα πλαίσια της εντολής από την διάσκεψη των προέδρων των Εθνικών Κοινοβουλίων το, ε, η Βελγική Βουλή των Αντιπροσώπων θα εμπλουτίσει με νέες προτάσεις τον όλο αυτό σχηματισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συναδελφοί. Έχουμε λιγότερο από μια ώρα για τη συζήτησή μας και έχω πάνω από 20 άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ λοιπόν να περιορίσετε τις παρεμβάσεις σας στα τρία λεπτά. Και θα δώσω αμέσως το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Αποθέσεων και Άμυνας της Γαλλικής Γερουσίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα στα γερμανικά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπροκ. Ε, τον ευχαριστώ για τα λόγια του. Έχουμε καταλάβει τις προθέσεις, είναι ξεκάθαρο ε, στα γερμανικά, αλλά θα καταλάβετε ότι δεν συμμεριζόμαστε απολύτω στη δική σας άποψη. Στα γαλλικά τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Βέλγο συνάδελφο για αυτά που μας είπε, διότι ε, και ευχαριστώ τη Βελγική Βουλή για τις προσ... το Βελγικό Κοινοβούλιο για τις προσπάθειές του. Στη κοινοβουλευτική συνέλευση της ΔΕΕ είναι το μόνο θεσμοθετημένο όργανο που επιτρέπει στη κοινοβούλια των 27 κρατών μελών να συνεδριάζουν με οργανωμένο τρόπο για να συζητούν από κοινού τα θέματα ευρωπαϊκής άμυνας. Οι κυβερνήσεις των 10 κρατών μελών της ε, ΔΕΕ ήταν 10, αποφάσισαν να θέσουν τέρμα στις ε, δραστηριότητες τους στον ερχόμενο Ιουλίου, τον ερχόμενο Ιούλιο, όπως αναφέρθηκε από τον προηγούμενο μιλητή. Δεν μπορούμε ωστόσο να προχωρήσουμε σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα που βρίσκεται ε, στο κέντρο της εθνικής κυριαρχίας χωρίς δημοκρατική νομιμότητα, απόλυτη δημοκρατική νομιμότητα. Ένα έλεγχος που θα ασκείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μόνο δεν θα αρκούσε κατά την άποψη άποψή Θυμίζω ότι οι αποφάσεις σε ό,τι αφορά τα αμυντικά ζητήματα εξαρτώνται από, είναι, αποτελούν αρμοδιότητα ενδιαφερομένων κρατών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις εθνικές κυβερνήσεις. Εξάλλου, οι ε, εθνικοί βουλευτές, όπως είπατε και εσείς αγαπητοί φίλοι, εκείνοι που ψηφίζουν για τους προϋπολογι... αμυντικούς προϋπολογισμούς και αναλαμβάνουν την αποστολή ή όχι στατευμάτων σε μία σύραξη. Εμείς στη Γαλλική Γερουσία ομόφωνα, το τονίζω αυτό, ομόφωνα αποφασίσαμε ότι η κατάργηση της συνέλευσης της ΔΕΕ θα έπρεπε να καλυφθεί από ένα οργανισμό στον οποίο να συμμετέχουν ε, βουλευτές ε, ερμόδιοι για τα θέματα άμυνας των 27 κρατών μελών. Σκεφτήκαμε να ακολουθήσουμε το πρότυπο της ΚΟΖΑΚ που είναι ένας οργανισμός που αναγνωρίζει τις συνθήκες και έχει ως εκ τούτου κάποια στοιχεία συνέχειας. Υπάρχει ένα άλλο πλεονέκτημα περιλαμβάνει εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αποτέλεσμα να μπορούν να συνεργάζονται οι εθνικοί και οι ευρωπαϊκοί βουλευτέ στα πλαίσια αυτού του οργάνου. Το πρωτόκολλο στη συνθήκη τη Λισαβόνας ορίζει ότι η ΚΟΖΑΚ μπορεί να οργανώνει διακοινοβουλευτικές διασκέψεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα για να συζητήσει θέματα εξωτερική πολιτική και κοινή ασφάλεια και άμυνα αφετέρου. Θα ήταν λοιπόν δυνατό πάνω σε αυτή τη βάση να, γίνουν, να οργανώνονται συνεδριάσεις τύπου ΚΟΖΑΚ στις οποίες θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των Επιτροπών Άμυνας των Εθνικών Κοινοβουλίων. Στόχος πρέπει να είναι να βρεθεί μια διαδικασία που θα εξασφαλίζει τη συνέχεια στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την εξέταση από τα κοινοβούλια των θεμάτων της άμυνας. Πρέπει να υπάρξει ένα σύνδεσμος ανάμεσα στα κοινοβούλια και την Ευρώπη της άμυνας. Πιστεύουμε ότι η παρούσα κατάσταση δεν επιτρέπει στους βουλευτές να παίξουν πλήρως το ρόλο τους. Γι' αυτό πρέπει να ε, ε, συμβάλλουμε στην διαμόρφωση καλύτερων συνθήκων. Η καλύτερη νήση θα είναι ο συνδυασμός των διαφόρων μορφών παρακολούθησης και ελέγχων νομιμότητας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ρόμπερτ Βόλτερ από τη Βουλή των Κοινοτήτων ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ αυτό που θυμήσατε ότι είμαι και πρόεδρος της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιος είπε ότι υπεξαιρέσαμε τις προνομίες το Μάρτιο διότι δεν είχαμε τον τίτλο και την εξουσιοδότηση να ασκούμε πάνω στην ΕΠΑ τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 12 νυν πρώην μέλη της συνέλευσης σήμερα και δύο πρώην πρόεδροι της Δυτικοευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης οι οποίοι θα επιβεβαιώσουν αυτά τα οποία σας λέω. Πρόεδρε, όπως ε, τονίστηκε, έχουν γίνει διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες συνεχίζονται αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι αυτό που οδηγεί τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι η άποψη που τονίστηκε ε, από τους προηγούμενους ομιλητές ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια και Εθνικές Κυβερνήσεις είναι εκείνα που ε, ε, αναπτύσσουν τις, τα στρατεύματά μας πληρώνουν τα έξοδά τους, αποφασίζουν πώς θα εξοπλιστούν οι ένοπλες δυνάμεις. Μιλάμε για διακυβερνητικές πολιτικές, όπως άλλωστε αναφέρεται και στις συνθήκες της Λισαβόνας. Εκείνοι οι οποίοι ε, εξέτασαν τα θέματα αυτά στα πλαίσια των αρμοδίων επιτροπών και επεξεργάστηκαν τις προτάσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων διαπίστωσαν ότι υπάρχουν αφενός εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να δημιουργήσουν ή να, να διατηρήσουν, να επαναδημιουργήσουν μια κοινοβουλευτική συνάλευση ενώ άλλοι λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα τέτοια και να αφήσουμε τα πάντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα στο οποίο ε, αναφέρθηκε στο άρθρο 90 του ψηφίσματος αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο το υπερεθνικό ε, όργανο που καλείται να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο για τις πολιτικές άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι εκπρόσωποι των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων ίσως δεν συμφωνήσουν με αυτό και θα, και θα ήθελα να επικρατήσει και να ευρεθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο. Όπως είπε ο συνάδελφο που μόλις μίλησε από τη Γαλλία, υπάρχει σκέψη δημιουργίας μιας ενός οργανισμού τύπου COSAC με τη συμμετοχή ή στη συμμετοχή όλων των, Ευρωπαϊκών, των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο χωρίς μόνιμη έδρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι μια λύση που θα επιτρέψει στα μέλη του, που θα ε, σημαίνει ότι θα, θα, τα, οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων θα έρχονται να ακούσουν ορισμένα πράγματα χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ουσιαστικό κοινοβουλευτικό όλογχο. Εγώ θα προτιμώ τη λύση της μόνιμης διάσκεψης με εκπροσώπηση των Εθνικών Κοινοβουλίων που θα συνεδριάζουν σε ολομέλεια δύο φορές το χρόνο και θα έχουν και άλλες συνεδριάσεις και θα υποστηρίζονται από μια μικρή γραμματεία και θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ως εθνικοί βουλευτές δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρόλο που η ΕΠΑ είναι, έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα. Εδώ στις Βρυξέλλες έχει δημιουργήσει διάφορες θεσμικές δομές που απαιτούν και αυτές κοινοβουλευτικό έλεγχο στο κατάλληλο επίπεδο, που είναι το επίπεδο των εθνικών κοινοβουλίων, των εθνικών βουλευτών, το Συμβούλιο, η ΚΟΠΣ, η Στρατιωτική Επιτροπή, το Στρατιωτικό και Αμυντικό Προσωπικό, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Καλό λοιπόν του εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων να μην ξεχνάνε τον ουσιαστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η συνέλευση τη Δικοπρακτική Ένωση για τόσα χρόνια και ελπίζω ότι ο οργανισμό που θα την ταδεχθεί θα συνεχίσει το έργο τη. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε μόλις τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της ΔΕΕ, που είναι το αρμόδιο όργανο για θέματα ασφαλείας, πρέπει να του πω ότι θα πρέπει να αποτίσουμε ένα φόρο τιμή στη συνέλευσή του για την ποιότητα των εργασιών του οργάνου αυτού από την ίδρυσή του. Κάποιος είπε προηγουμένως ότι οι εκθέσεις δεν ενδιαφέρουν κανένα. Δεν ισχύει αυτό. Σας προκαλώ να τις διαβάσετε και να δείτε τι επίπεδο είναι. Στη συνέχεια, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ρεαλιστές, πραγματιστές για το κοινοβουλευτικό έλεγχο. Λοιπόν, προπολογισμός. Ποιος το ελέγχει ε, τα εθνικά κοινοβούλια. Το ΚΑΒΕΑΤ, το κράτη-μέλη επίσης και τα εθνικά κοινοβούλια για τις ρήτρες τις διάφορες. Ε, τις αμυντικές δαπάνες, προμήθειες, σχεδιασμό, ε, βράχη πρόθεσμα, μέσο, μακροπρόθεσμα και πάλι τα εθνικά κοινοβούλια. πυρηνικά δύο είναι τα κράτη-μέλη που έχουν πυρηνικά. Δεν είμαι βέβαιος αν έχουν λόγο καν τα κοινοβούλια των δύο αυτών κρατών για τα πυρηνικά. Πάντω οι υπόλοιπε 25 χώρε δεν έχουν κανένα λόγο απολύτω για την πυρηνική ε, δύναμη. Οπότε υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα. Ας κάνουμε μια απογραφή λοιπόν, χωρίς καμία συγκατάβαση και σας προτείνω να επιφορτιστεί ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εσείς ο ίδιος και κάποιοι άλλοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια για να κάνουμε αυτή την απογραφή των ελλημάτων και να δούμε τι προτάσεις μπορούμε να υποβάλουμε σε εύθετο χρόνο και σε επόμενη συνεδρίαση για να είμαστε βέβαιοι ότι συζητούμε όλοι για το ίδιο πράγμα. Παρατήρηση δεύτερη. Ο κ. Ντουκάρμ πρότεινε πολλές φόρμουλες και πραγματικά θέλω να τον συγχαρώ για την ποιότητα της παρέμβασής τους, ε, αλλά παραμένουν μεγάλες ελλείψεις. Κόζακ, ας μην γελιόμαστε. Πολύ συχνά είναι 27 μονόλογοι και έρχεται να προσθεθεί και ένας 28ος. 27 εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, είναι σαν βαζάκι ο ένας δίπλα στον άλλον και κάθονται αμήλυτοι, ακίνητοι και ακούνε τους μονολόγους. Ε, αυτό δεν είναι συνέλευση. Η διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Ε, κατά γενικό κανόνα είναι εκπροσώπηση των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών των 27. Αυτό είναι άραγε αρκετά δημοκρατικό. Εγώ παραμένω στην άποψη που λέει όχι. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν και μια διαφοροποίηση στη σύνθεση αυτών των συνελεύσεων και θέλω να σταματήσω εδώ για να σεβαστώ και το τρίλεπτό μου. Αλλά ας προσπαθήσουμε, και αυτή είναι η πρότασή μου καθώς και το συμπέρασμά μου, να είμαστε ρεαλιστέ νυφάλοι, για να έχουμε την καλύτερη και την ίδια όλη ανάγνωση. Για να ξέρουμε ότι όλοι συζητάμε για το ίδιο ακριβώ πράγμα. Η κυρία Μέλγκαρτ, που είναι πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από το Κοινοβούλιο της Δανία. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και σα ευχαριστώ διότι λάβατε, αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία διοργάνωσης αυτής της συνάντησης, έτσι ώστε να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συναδέλφων για τη μελλοντική μας συνεργασία και τη μορφή που θα προσλάβει αυτή η συνεργασία. Όταν μιλάμε για την ΕΠΑ και γενικότερα για θέματα ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ε, Βουλή της Δανίας συζητάμε αυτό το ζήτημα και η Βουλή μας ασχολείται με τη διεύρυνση της συνεργασίας όταν μιλάμε για θέματα που άπτονται της άμυνας και της ασφάλειας δυνάμει του πρωτοκόλου 1 της συνθήκης της Λισαβόνας. Θεωρούμε ότι ο έλεγχος και η εποπτεία της νομιμότητας είναι κάτι που αφορά τα εθνικά κοινοβούλια. Το σημείο εκκίνησης για μας είναι ότι υποστηρίζουμε το House of Lords στην πρότασή του και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει, οι Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να συνέρχονται οπωσδήποτε μία φορά το εξάμεινο. Θα είχαμε έξι εκπροσώπους ανά κοινοβούλιο και η Προεδρία των Επιτροπών Ασφάλειας και Άμυνας είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό. Θεωρούμε ότι για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σχήμα, θεωρούμε ότι η Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να, ε, στην Επιτροπή αυτή θα πρέπει να υπάρχει ε, ισοψηφία. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει σωστή εκπροσώπηση σε αυτές τις συναντήσεις. Επίσης, θα θέλαμε να υπάρχει πολιτική ευθύνη για τον προγραμματισμό και θα πρέπει η Τρόικα να αποφασίσει και η ΚΟΖΑΚ θα πρέπει να μας βοηθήσει ως προς την ε, ε, γραμματιακή υποστήριξη στις Βρυξέλλες. Η Βουλή της Δανίας προσδίδει μεγάλη σημασία στην ΚΟΖΑΚ όταν μιλάμε για την οργάνωση αυτών των διακοινοβουλευτικών διασκέψεων. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να συσταθεί μία νέα γραμματιακή δομή για να υποβοηθήσει το έργο αυτής της διακοινοβουλευτικής διάσκεψης. Εγώ ως ε, πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών, ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από πλευράς Δανίας. Θα ήθελα να εκπροσωπηθώ, αλλά δεν θα ε, μεταβαίνω εγώ κάθε φορά. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια νέα μορφή συνεργασίας δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Σερνό, από την Πορτογαλία. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ε, μιλήσω για θέματα άμυνας και ασφάλειας και ευχαριστώ τον πρόεδρο της Υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας που ε, προέβλεψε να συγκαλέσει αυτή την συνάντηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Έλμαρ Μπρόκ για την εισήγησή του καθώς και τον εκπρόσωπο της Βελγικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι στον τομέα της πολιτικής στα πλαίσια των νέων αρμοδιοτήτων της συνθήκης της Λισαβόνας θα πρέπει να δημιουργήσουμε ε, ένα μηχανισμό εποπτείας και ελέγχου αυτών των αρμοδιοτήτων και αυτός ο έλεγχος έχει δύο πλευρές. Αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική και τις νέες αρμοδιότητες που εμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο και μια δεύτερη διάσταση αφορά τις ειδικέ αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να συνεργαστούν στον τομέα της χρηματοδότησης, του εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων και της μετάβασης ή απόσπασης των ενόπλων δυνάμεων όπου χρειάζεται. Αυτό αφορά και τον, ε, έλεγχο, τον γενικότερο έλεγχο της νομιμότητας. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που διαμορφώνονται πλέον. Είχαμε, υπήρχε πολιτική ε, νομιμότητα μέσα στα πλαίσια της ε, Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, όμως η δε που εξαρτάται από ε, από μορφές κοινοβουλευτικού ελέγχου διαλύεται. Γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει και ε, έλεγχος από πλευράς Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Και γι' αυτό υπάρχουν ε, διάφορες νέες μορφές ελέγχου της νομιμότητας που προβλέπονται δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Άρα θα πώς διαμορφώνεται αυτός ο έλεγχος. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πείρα του παρελθόντος και της ΔΕΕ και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που προείπαν οι εκπρόσωποι της, ε, του, της Βελικής Βουλής των Αντιπροσώπων ή ο Γάλλος εκπρόσωπος. Θα πρέπει να υπάρχει όμως ένας έλεγχος, εθνικός έλεγχος νομιμότητας είτε στα πλαίσια της ΕΠΑ είτε της ΚΕΠΑ. Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται μόνιμα ή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εδώ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα ήθελα να τονίσω και μία άλλη πλευρά του ζητήματος. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 27 κρατών μελών, θα πρέπει να ε, εξάρουμε και το ρόλο των επιτροπών εξωτερικών υποθέσεων και των επιτροπών, εθνικών επιτροπών άμυνας και ασφάλειας. Γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 21 κράτη-μέλη συμμετέχουν και στις δομές, στη δομή του ΝΑΤΟ από τα 27 κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς διαμορφώνεται ο ρόλος αυτών των χωρών και να δούμε πώς θα υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο συνεργασίας και των 27. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα δράσουν και οι ΚΟΦΑΚ και οι ΚΟΝΤΑΚ στο μέλλον. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πείρα μας στα πλαίσια της ε, Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουμε μία μικρή και ευέλικτη γραμματεία, περιορισμένη γραμματεία και να χρησιμοποιήσουμε την ε, πείρα του παρελθόντος με βάση τα, ε, την, την πείρα και τα δρόμενα στην Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε μελλοντικά και την ΕΠΑ και την ΚΕΠΑ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Σας θυμίζουμε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Δεν πρέπει να ξεπερνάτε τα τρία λεφτά για να μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο όσοι τον ζήτησαν. Θα... Σας ειδοποιώ με το σφυρί μου ότι ο χρόνος σας τελείωσε. Μόλις ολοκληρώσετε τα τρία λεπτά. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ. Και εγώ νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι ύψης της σημασίας διότι θα πρέπει να δώσουμε μία σωστή διάρθρωση στην ε, εποπτεία της νομιμότητας που εμπίπτει και αφορά τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνάμη της συνθήκης της Λισαβόνας όπως ε, προϋπόθηκε. Συμφωνώ με τον κύριο Αρναούτ ε, σε σχέση με την διάρθρωση αυτή και πώς θα πρέπει να συνεχιστεί μετά τη λήξη των εργασιών της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι από τη μία πλευρά Δεν πρέπει να είμαστε υπέρμαχοι του γεγονότος ότι η υποεπιτροπή θα πρέπει να μετατραπεί σε επιτροπή που να ασχολείται με θέματα άμυνας και ασφάλειας και να διαδραματίσει το ρόλο που διαδραματίζει η ΑΦΕΤ. να αφορά κάτι το μελλοντικό, αλλά νομίζω ότι η υποεπιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να είναι υποεπιτροπή να συνεργάζεται με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, διότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας έχει μία διαφορετική διάρθρωση και δομή. Και αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτό το σχήμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε κάπως ευέλικτοι σε αυτή τη διάρθρωση. Δεν θα πρέπει να ε, έχουμε μηχανισμούς που να είναι ανέλικτοι και που καθιστούν την διάδραση κενή περιεχομένου. Όπως είπε και ο Σνάφος Γκέρενς, η Κόζακ ίσως ε, απαρτίζεται από 27 συν ένα μονολόγους, δηλαδή 28 μονολόγους, κάτι το οποίο δεν θα ήταν ε, σκόπιμο. Θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική ε, διάδραση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ κοινοβουλίων. Γι' αυτό είμαι υπέρ μιας λύσης που πρότεινε και η εκπρόσωπος της Δανίας, δηλαδή να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων, μια πραγματική διάδραση και όχι μία ε, ανέλικτη ή ειδική γραμματεία. Γιατί σε αυτή την ε, περίοδο ε, κρίσης δεν θα γινόταν κατανοητό από τους πολίτες μας ε, αυτή η κατασπατάληση χρήματος για τη σύσταση μιας νέας γραμματείας. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια σωστή συνέχεια και διάδραση με τα εθνικά κοινοβούλια. Έτσι, όλοι οι βουλευτές θα συμμετείχαν σε αυτό το διάλογο με στα πλαίσια των Εθνικών Επιτροπών Άμυνας και Ασφάλειας και Εθνικών Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βρετός, παρακαλώ, πρόεδρος της ε, Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να θυμηθούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι για τις αποφάσεις της κοινής ευρωπαϊκής και αμυντικής πολιτικής, ε, της κοινής Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας χρειάζεται ομοφωνία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας διακυβερνητικός χαρακτήρας, άρα ο ρόλος των ελληνικών κοινοβουλίων είναι κυρίαρχος. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει περισσότερες αρμοδιότητες στα θέματα της άμυνας. Αλλά τα ελληνικά κοινοβούλια παραμένουν εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντικά. Και με αυτή την έννοια θα συμφωνήσω με, πάρα... με τον Γάλλο συνάδελφο και με άλλους συναδέλφους που μίλησαν πάνω σε αυτό. Δεύτερο, ε, άκουσα τον κύριο Μπροκ και λυπάμαι γιατί διαφωνώ σε αρκετά σημεία με αυτόν. Ε, πρώτον, ε, το, ο κύριος Μπροκ, αν κατάλαβα καλά, θέλει, προτείνει να έχουμε να μαζευόμαστε εδώ οι πρόεδροι των επιτροπών, προσέξτε, οι πρόεδροι των επιτροπών των Ελληνικών Κοινοβουλίων με την επιτροπή σας και να αποφασίζουμε. Αυτό είναι κατά την άποψή μου υποτιμητικό για τα ελληνικά κοινοβούλια και αναποτελεσματικό. Από όπου και σπου μόνο οι πρόεδροι θα συμμετέχουν και εδώ ολόκληρη η επιτροπή θα είναι που θα συζητάει τα θέματα αυτά. Δεύτερο, μου έκανε εντύπωση επίση από τον κύριο Μπρόκ ότι είπε ότι ε, δεν χρειάζονται οι μελέτες, ε, δεν χρειάζονται οι, οι εισηγήσει, δεν χρειάζονται οι γραμματείες κλπ. Φανταστείτε εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε γραμματιακή υποστήριξη καλή, αν δεν είχε εισηγήσει, αν δεν είχε εισηγητέ. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμά του. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Τρίτον, ήθελα εδώ να πω ότι η Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αδικηθεί από, την, από το ε, Ευρωκοινοβούλιο αλλά και γενικότερα από, την, από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει κάνει πολύ σπουδαίο έργο, πολύ σημαντικό και μακάρι να το είχαν παρακολουθήσει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δική σας Επιτροπή. Δεν το έκαναν. Και εδώ έχουμε σημαντικά πρόσωπα τα οποία ξέρουν, έχω μπροστά μου, τυχαία το βλέπω, τον κύριο Ντεντεκέρ, επειδή είναι μέλος και πρώην πρόεδρος της Γερουσίας. Μεγάλη συμβολή, μεγάλη προσφορά. Εσείς Δυστυχώ, και λυπάμαι γι' αυτό, δεν καλέσατε τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης επισήμως να συμμετέχει σε έναν διάλογο ο οποίος κυρίω στον οποίο θα μπορούσε κυρίως να προσφέρει πάρα πολλά. Ε, τώρα, για να μην είμαι ε, ε, εντελώς αρνητικός, ήθελα να σας πω ότι η πρότασή μου είναι ότι πρέπει να γίνει ένα όργανο που να, είναι, να έχει αναλογική ε, συνεισφορά από τα κράτη-μέλη, από βουλευτές. δεύτερον, να υπάρχει μια ολιγομελής γραμματεία, όχι μεγάλη. Και αυτό που ε, άκουσα προηγουμένω από την ε, συνάδελφό μα του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν μιλάμε για πολλά χρήματα. Δεν μιλάμε για σπατάλη. Μιλάμε για μικρή γραμματεία η οποία θα μα υποστηρίζει. Και με την, να έχουμε επιτροπέ και εισηγητέ, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συνθέσουν μια σοβαρή αντίληψη πάνω στα θέματα τη κοινή πολιτική ασφαλεία και άμυνας. Και ε, θα ήθελα να σα πω ότι τα, πρέπει, αν ο προπολογισμό, ο οποίο είναι μικρό κατά την άποψή μου, θεωρηθεί πολύ μεγάλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, α αποφασίσουν τα ελληνικά κοινοβούλια να το κάνουν αυτό. Οφείλουν να το κάνουν. Διαφορετικά δεν μπορούμε να εκφραστούμε. Διαφορετικά δεν μπορούμε να περάσουμε τα μηνύματά μα προ τι δικέ μα επιτροπέ και στα δικά μα ε, κοινοβούλια. Ε, νομίζω ότι από του ε, συναδέλφου μα υπόθηκαν πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Για την Κόζακ, εγώ προσωπικά δεν διαφωνώ να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά έτσι όπω είναι η Κόζακ δεν κάνει. Δεν κάνει, διότι δεν είναι αποτελεσματική. Ε, κάναμε μεγάλε προσπάθειε, θυμάμαι, ήμουν κάποτε προεδρεύω τη Κόζακ και καταφέραμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, δηλαδή να έχει μια στοιχειώδη γραμματεία και να παίρνει μια αποφάσει. Παρ' όλα αυτά όμω θα σα θα σας το πω καθαρά ότι δεν, η Κόζακ δεν είναι αποτελεσματική γιατί δεν θέλουν οι βουλευτέ που συμμετέχουν από το Ευρωκοινοβούλιο εκεί να την βοηθήσουν να είναι αποτελεσματική. Άρα λοιπόν προτείνω να γίνει η συνέλευση, αυτή την οποία ε, έχουν προτείνει και άλλοι συνάδελφοι, να είναι ένα όργανο πολύ καλύτερο από την ΚΟΖΑΚ και ίσως υποδέστερο από την Συγγνώμη, υποχρεωμένο να σα διακόψω. Συνάδελφοι, ο χρόνο μα είναι περιορισμένο. Υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να πάρουν τον λόγο και θα ήθελα να έχουν τη δυνατότητα όλοι να μιλήσουν. Παρακαλώ λοιπόν να μην ξεπερνάτε τα τρία λεπτά. Ο κύριος Φόρσλουντ, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Σουηδικής Βουλής. Θα προσπαθήσω, Πρόεδρε, να τηρήσω τα τρία λεπτά. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη φιλοξενία του και δεύτερον θέλω να θυμίσω ότι στις παραγράφους για την κοινή ε, πολιτική άμυνας και ασφάλειας, την ΕΠΑ, παράγραφοι 6 και 7 από τα συμπεράσματα της Επιτροπής των Προέδρων στη Στοκχόλμη, οι πρόεδροι των κοινοβουλίων είπαν, λόγω της ειδική φύσης της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πρόεδροι υπογραμμίζουν τον θεμελιώδη ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στη μελλοντική διαδικασία ελέγχου της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής. 7. Οι πρόεδροι ζήτησαν την περχόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία στην επόμενη συνάντηση της ε, ε διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε για μια φορά ακόμη ότι οι πρόεδροι υπογράμμισαν τον σημαντικό ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στα πλαίσια της μελλοντική διαδικασίας ελέγχου. Είμαστε ευγνώμονες που η Προεδρία θα δώσει συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση, πάνω σε αυτή τη βάση, με βάση τις αποφάσεις που έλαβαν οι εκπρόσωποι της Εστονίας της Λιθουανίας και άλλων χωρών πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα για την κοινοβουλευτική συνεργασία υπό την αιγίδα των Εθνικών Κοινοβουλίων χρησιμοποιώντας την τρέχουσα δομή, την υφιστάμενη δομή ως βάση. Τούτου λεχθέντος θέλω να υπογραμμίσω το ενδιαφέρον που έχει επιδείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τον βουλευτικό έλεγχο της ΕΠΑ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση ενός τέτοιου ελέγχου. Αναφέρουμε επίσης ότι, πρέπει, ε, ότι, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προσωπείται στην ΚΟΦΑΚ και στην ΚΟΝΤΑΚ και χαιρετίζουμε τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη λειτουργία αυτών των δύο επιτροπών. Ευχαριστώ. Σας συγχαίρω για την πειθαρχία σας. Είστε ο πρώτος που δεν ξεπέρασε τα τρία λεπτά. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η έκθεση Μπροκ για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ήταν επιτυχία από πλευράς Κοινοβουλίου και σε ε, περίοδους κρίσης δεν ε, ασχολήθηκαν πάρα πολύ οι ηγέτες μας τότε ε, γιατί ήταν αποσπασμένοι αλλού. Ενώ η έκθεση Μπροκ εξασφαλίζει και πολλά δικαιώματα όπως είπε, να έρχονται και στην Επιτροπή Εξωτερικών οι πρέσβει και οι πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πριν ε, αναλάβουν τα καθήκοντά του. Τα εθνικά κοινοβούλια δεν ε, απολαμβάνουν όλοι αυτών των δικαιωμάτων. Η δική μου ομάδα θεωρεί ότι οι εθνικές κυβερνήσει και οι εθνικές βουλές είναι θεμελιώδεις για την ασφάλεια και την άμυνα στην Ένωση. Και μόνο οι εθνικοί βουλευτές αποφασίζουν ε, αν θα στείλουν στρατεύματα σε κάποιο πόλεμο γιατί οι φαντάροι μας σκοτώνονται για τα κράτη μας, όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι αφορά τιμή στο συνάδελφο Μπομπ Γόλτερ για το ρόλο του ε, ως πρόεδρο της συνέλευσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό το όργανο θα διαλυθεί του χρόνου και πρέπει από κάτι να αντικατασταθεί. Δεν μπορούν ε, και οι εθνικοί βουλευτέ να αποκλείσουν τελείω του ευρωβουλευτέ από τι αποφάσει Γιατί για τις πολιτικές αποστολές ε, χρηματοδοτούνται, α πούμε το Γιούλεξ στο Κόσοβο, οι υπάλληλοι από κοινοτικά κονδύλια και είναι ε, ε, αυτές οι πολιτικές ε, αποστολές η πλειονότητα των αποστολών στην ΕΠΑ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια νέα συνεργασία, συνεργασία και όχι αντιπαλότητα με τα εθνικά κοινοβούλια. σε μια εξάμεινη διάσκεψη, προτιμώ το διάσκεψη παρά το συνέλευση γιατί δεν έχει νομική βάση. Ούτε θέλω να διαχωριστούν οι ΚΕΠΑ από την ΕΠΑ γιατί τόσο πολύ επικαλύπτονται. Ξέρω ότι υπάρχει και κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ χωρίς νομική πάντα βάση στο Βόρειο Ατλαντικό Σύμφωνο. δεν συμμετέχουν πάντα πολλοί βουλευτέ ούτε ευρωβουλευτέ. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν πρόεδροι, συμπρόεδροι, στάθμιση ανάλογα με την Εθνική Βουλή και πάλι αυτό ε, παραμένει να συζητηθεί. Εγώ προτείνω ε, και προτιμώ η γραμματεία να είναι ε, από του εθνικού προπολογισμού και να συνεδριάζει το Συμβούλιο και όχι σε Κοινοβούλιο και να υπάρχει και ένα είδος ε, εναλλαγής. Δεν θα σας εκπλήξει, διαφωνώ με την πρόταση συμβολή στο Λόρδο, Έξι βουλευτές μόνο στην ΚΟΦΑΚ και ΚΟΝΤΑΚ χωρίς δική μας εκπροσώπηση. Και θα είναι κάποιος τελείως παράλογος εκπρόσωπος ε, και θα αποκλείονται από το ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόσφατα κάναμε μια συζήτηση πάρα πολύ εκρινή και η δική μας αντιπροσωπεία συμφωνούσε σε γενικές γραμμές με μένα. Και ένας γνωστός ευρωσκεπτικιστής χρειάστηκε τους ευρωβουλευτές γιατί ε, παραδέχτηκε, ε, παρακαλώ, ότι οι ευρωβουλευτές είναι οι μόνοι που καταλαβαίνουν το λαβύρινθο και τους δεδάλους εδώ των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ντεντεκέρα, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και αμήνη της Βελγικής Γερουσίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και ευχαριστώ ειδικότερα την Υποεπιτροπή που οργάνωσε τη σημερινή μας συνάντηση η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική κατά την άποψή μου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνεδριάζουμε σήμερα ε, συνδέονται Βεβαίω με την εξέλιξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη θέση της συνθήκη Λισαβόνα, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την καταγγελία της τοποποιημένης συνθήκης των Βρυξελών. Αυτό που θα ήταν ωστόσο υπερβολικό και λυπηρό θα ήταν να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια ουσιαστική πρόοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συνθήκη της Λισαβόνα, η οποία όμως δεν πρέπει να δημιουργήσει δημοκρατικό έλλειμμα σε έναν τομέα τόσο σημαντικό όπως είναι ο τομέας της άμυνας και της ασφάλειας. Κάτι που μπορεί φοβάμαι να συμβεί αν συνεχίσουμε να ε, ενισχύουμε μία αντιπαλότητα μεταξύ των Ευρωπαίων Ευρωβουλευτών, ε, των Ευρωβουλευτών αφενών και των Εθνικών Βουλευτών. Ακούγοντα τον κύριο Μπρόκ, οι πολιτικέ αποστολέ είναι πολυπληθέστερε από τι στρατιωτικέ. Οπότε, χωρί να σημαίνει αυτό ότι μειώνεται ο δραματικό, τραγικό χαρακτήρα των στρατιωτικών αποστολών και πόσο δύσκολε είναι οι αποφάσει που πρέπει να ληφθούν για να σταλούν άνδρε ε, φαντάρι σε, να λάβουν μέρο σε στρατιωτικέ αποστολέ η κοινοβουλευτική συνέλευση της ΔΕΕ, η οποία θα εξαφανιστεί, προσέφερε πάρα πολύ σημαντικές υπηρεσίες στους ε, βουλευτές επί 60 χρόνια, βοηθώντας τους να αποκτήσουν μία ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή θεώρηση, ξεφεύγοντας από το στενό εθνικό πλαίσιο το οποίο όταν θέλει κανείς να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας δεν είναι κάτι το χρήσιμο. Επικαλούμε λοιπόν τη συνθήκη. Η συνθήκη στο άρθρο 9 μας λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια ορίζουν από κοινού τη συνεργασία τους, πρώτο σημείο, και το άρθρο 10 κατόπιν λέει ότι από κοινού μπορούν να συστήνουν όργανα εξειδικευμένα για τα θέματα τα οποία κρίνουν χρήσιμα και σκόπιμα. Σας ερωτώ λοιπόν και απευθύνομαι στους ευρωβουλευτές και στους εθνικούς βουλευτές ζητώντας τους να εφαρμόσουν τη συνθήκη και να αποφασίσουν θα συνεργαστούμε από κοινού οι εθνικοί βουλευτές και οι ευρωβουλευτές σε μια μόνιμη διακοινοβουλευτική συνέλευση. Ποιο θα είναι το πλεονέκτημα? Ότι κάθε χρόνο θα ακούμε μια έκθεση του Συμβουλίου για όλα αυτά τα θέματα και θα αναπτύσσουμε διάλογο με το Συμβούλιο. Και ισχυρίζομαι και είμαι μάλιστα απόλυτα πεπισμένος ότι αν δημιουργήσουμε μια κοινή συνέλευση μεταξύ Ευρωπαίων και Εθνικών Βουλευτών, οι Ευρωπαίοι Βουλευτές και είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποκομίσουν, θα αποκομίσουν ε, σημαντικά στοιχεία, σημαντικά στοιχεία, σημαντική ενημέρωση και αυτό ισχύει από τους εθνικούς βουλευτές. Αντίστοιχα δε οι εθνικοί βουλευτές θα ωφεληθούν από την επαφή και τη συνεργασία με τους ευρωβουλευτές Υπάρχουν οι δομές, υπάρχει γραμματεία, ε, στην, ε, στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει γραμματεία στα Εθνικά Κοινοβούλια που θα μπορούν να συνεργαστούν, υπάρχουν οι αντίστοιχε επιτροπές που και αυτές θα συνεργάζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε όλοι οι βουλευτές όταν χρειάζεται να αποφασίσουν την αποστολή στρατευμάτων και ψηφίζουν το σχετικό προπολογισμό να το κάνουν για το καλό της δικής τους χώρας αλλά και για το καλό του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης membre de la Commission des Affaires étrangères. Ο εκπρόσωπος τώρα της Φιλανδικής Βουλής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, ε, ε τους κύριους Μπροκ και ε, Ντουκάρμ για την ε, συνδρομή τους. Θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα συνεχιστεί αυτός ο διάλογος για θέματα ασφάλειας και άμυνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη Φιλανδία η ΕΠΑ είναι ύψη της σημασίας και θεωρώ ότι αυτό ισχύει και για τις άλλες χώρες που δεν συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ. Στην Φιλανδία έχουμε ένα ενδελεχές σύστημα εποπτείας της νομιμότητας που βασίζεται στο Σύνταγμα. Γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε την ε, προσοχή μας στην εποπτεία σε εθνικό επίπεδο, γιατί εκεί είναι ελληματική. Θεωρούμε επίσης ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συνεχίσουν το διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Θα πρέπει δηλαδή να είναι μία προσθέμενη αξία ως προς την εργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνδράμει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εργασία των Εθνικών. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπορούν και μέλη που δεν συμμετέχουν στην Ευρω... Ε, κράτη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη δομή. Επίσης, μας ενδιαφέρει η, η ενίσχυση των ευρωπαϊκών ε, δομών και εκτός ΝΑΤΟ. Ο πιο ε, πρακτικός τρόπος και εποφελής από πλευράς χαμηλών δαπανών ε, θα ήταν να δούμε πώς μπορεί να οριστεί αυτή η συνδρομή από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επειδή πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ποιότητα, θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις από το νέο αυτό ε, σώμα. Στα πλαίσια της ε, διακοινοβουλευτικής διακοινοβουλευτικές συνεργασίας θα πρέπει να υπάρχει ε, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μια πραγματική συζήτηση και ανοιχτή συμμετοχή όλων και αυτών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να έχουμε μία σωστή σχέση κόστους-οφελίας, να μην έχουμε μία επιβαρημένη γραμματεία και ανέλικτη γραμματεία και να συμμετέχουν όλες οι χώρες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθός τους. Σας ευχαριστώ. Ο Άντριου Ντάφ έχει το λόγο. Πρόεδρε. Το θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα πρέπει να διέπεται από ένα ερώτημα. Πού βρίσκεται η εξουσία. Το θέμα δεν είναι η εκπεριτροπής προεδρία. Δεν έχουν εκείνη την εξουσία. Είναι η μόνιμη προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Μία λύση τύπου Κοζάκ βασίζεται στην παραδοχή ότι η εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου διαδραματίζει ακόμα ρόλο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μία λύση τύπου Κόζακ σε μεγάλο βαθμό υποεκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν μειώσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν είμαστε συνεπείς στη λογική, στο πνεύμα δηλαδή της συνθήκης της Λισαβόνας. Η συνθήκη έρχεται να συμπληρώσει τη διακυβερνητική διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΚΕΠΑ και στην ΕΠΑ με μια, κοινοβουλευτική, με μια συγγνώμη, κοινοτική διάσταση. Η κάθε άστον που είναι και επίτροπος μπορεί να ε, προτείνει πολιτικές και το Συμβούλιο να αποφασίζει κατά ε, πλειοψηφία για τις πολιτικές αυτές. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν αντιλαμβάνονται ε, αυτό το θέμα. Τις λεπτές αποχρώσεις δηλαδή. Έχουμε τρεις κοινοβουλευτικές λειτουργίες την ξεχωριστή λειτουργία με το ιστορικό ρόλο και το κύρος που αναλογεί σε κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο. Είναι μία διάσταση. Απ' την άλλη έχουμε και πάλι μια ξεχωριστή διάσταση που είναι νέα, που είναι οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα πρέπει επίσης να υλοποιούνται στην πράξη αποτελεσματικά, αλλά και υπάρχει και μια τρίτη διάσταση που είναι η κοινή ε, σε συνεργασία λειτουργία για να αναζητήσουμε τι κοινό έχουμε. Όλα τα κράτη. Ποια είναι ας πούμε, η ανησυχία της Ευρώπης για την ασφάλεια και το μέλημά της. Και δική μας λοιπόν αποστολή σε αυτό το διακοινοβουλευτικό ε, τύπο συνεργασίας είναι πρώτα απ' όλα να καθορίσουμε αυτό το κοινό μας συμφέρον και στη συνέχεια να λάβουμε υπόψη και τις οικονομικές και τις πολιτικές ε, συνέπειες των ε, επιχειρησιακών αποφάσεων που προέρχονται από την ΚΕΠΑ και την ΕΠΑΑ. Νομίζω ότι είναι απλό αυτό το εγχείρημα και κανονικά δεν θα έπρεπε να μας υπερβαίνει κιόλα να μας ξεπερνάει. Θα μπορούσαμε να είμαστε σε θέση κανονικά να έχουμε μια ε, συνενετική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα και στο ε, διακοινοβουλευτικό διάλογο και συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φρουνζούλητσα, μέλος της Επιτροπής Αμήνης της Ρουμανικής Βουλής. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αυτός ο διακοινοβουλευτικός ε, διάλογος σε σχέση με την ΕΠΑ και την ΚΕΠΑ είναι ύψης της ε, σημασίας γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το διπλό δημοκρατικό έλλειμμα όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αρκετές εξουσίες λήψης αποφάσεων, αλλά πολύ καλές γνώσεις και ολοένα και ε, με γενθυμένο ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Αλλά τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν μεγάλες εξουσίες, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν ως προς τις απαιτήσεις λήψης αποφάσεων σε θέματα ΕΠΑ και ΚΕΠΑ. Μόνο με την κοινή δράση Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού θα μπορέσουμε να φτάσουμε στη δημοκρατική νομιμότητα που απαιτείται για την ΕΠΑ. Κυρίες και κύριοι, ένα από τα ε, ευαίσθητα ζητήματα είναι η διάλυση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με θέματα άμυνας και ασφάλειας. Από τη μία πλευρά το πέρασμα της ε, ΔΕΕ στη συνεργασία Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού σημαίνει ότι μπορούμε να επηρεάσουμε και τον προϋπολογισμό και τις ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Από την άλλη πλευρά, η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε θέματα λήψη αποφάσεων. Εφόσον όμως υπάρχει η ΚΟΖΑΚ, πιστεύω ότι θα μπορούσε να ασχοληθεί με θέματα άμυνας και ασφάλειας και όπως έγινε ήδη μια πρόταση εδώ, ένα σώμα που να μοιάζει με την ΚΟΖΑΚ θα μπορούσε να αντικαταστήσει την τελευταία. Η συνθήκη της Λισαβόνας μιλά για καλύτερη εποπτεία, αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να εξεύρουν τα κατάλληλα μέσα έτσι ώστε η διάταξη αυτή να μην παραμείνει ή να μην μετατραπεί σε χάρτινο τίγρη. Θα πρέπει να επέλθει μεγάλη βελτίωση. Σύμφωνα με τη συνθήκη, τα κράτη-μέλη μπορούν να λάβουν αυτοβούλως αποφάσεις σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Γι' αυτό μπορούν να επηρεάσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με συγχωρείτε, μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας μπορούμε με βάση τους υπάρχοντες μηχανισμούς να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Εφ' Ο διακοινοβουλευτικό διάλογος δεν προβάλλει μόνο την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, αλλά αποτελεί μέσο δημοκρατικού ελέγχου και εποπτείας των ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Από τη Βουλή των Λόρδων, ο κύριος Ρούπερ. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση συνδράμει στην συζήτηση της Στοκχόλμης το Μάιο και της Κόσα και τη συνάντηση της Κόσα και Κόφακ, καθώς και τη συνάντηση του Δεκεμβρίου που προανέφερε ο κύριος Μπρόχ που δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Έγιναν ήδη συζητήσεις και οι πρόεδροι των επιτροπών του, της Βουλής των Αντιπροσώπων ε, ήρθαν σε επαφή μαζί μου και μιλήσαμε για το έγγραφο που προέβαλε η Βουλή των Λόρδων. Χαίρομαι διότι υποστηρίχθηκε σήμερα. Βασιζόμαστε στο άρθρο 10 του πρωτοκόλου 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας που αναφέρει ότι η ΚΟΖΑΚ μπορεί να διοργανώσει διακοινοβουλευτικές διασκέψεις για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τις ΕΠΑ και ΚΕΠΑ. Το άρθρο 9 δεν δεσπόζει του 10 δεν επικρατεί του 10 και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η σημερινή συζήτηση με τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης θα πρέπει να προβάλλουμε την εργασία των ΚΟΦΑΚ και ΚΟΝΤΑΚ δηλαδή να δημιουργήσουμε μία διάρθρωση με έξι βουλευτές από κάθε κοινοβούλιο, ε, να πω να προσέλθουν και ε, πρόσωπα από τα διάφορα κόμματα ή τις επιτροπές όπως προανέφερε και η ε, Δανέζα βουλευτής. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και ο κύριος Τάνοκ είπε για ε, έξι εκπροσώπους από όλες τις πολιτικές ομάδες. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Δεν θα πρέπει να έχουμε μία ε, βαριά διάρθρωση, θα πρέπει να είναι πιο ανάλαφρη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν μπορούμε να σπαταλήσουμε τόσα χρήματα αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε μία συνέχεια ως προς τις γραμματιακές ε, υπηρεσίες και δομές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αξία αυτού του εγχειρήματος, διότι δεν θα πρέπει να έχουμε σωρία εκθέσεων. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι έμεσα και όχι άμεσα, δηλαδή ε, η εποπτεία θα πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που κατέχουν επαρκώς το θέμα και μπορούμε να το κάνουμε αυτό με μια ιδιαίτερα ανάλαφρη δομή. Ο κύριος Μπολτιέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση που δεν είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν. Και θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό με βάση καινοτόμα στοιχεία και να υπάρχει και μία αμοιβαία κατανόηση βεβαίως. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι τα εθνικά κοινοβούλια οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε σχέση με μια πολιτική που αποφασίζει το Συμβούλιο και ειδικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτά τα δεδομένα και να γνωρίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να ασκήσουν έλεγχο σε αυτή την νομιμότητα. Αυτό το οφείλουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες και θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το στοιχείο, που είναι ένα στοιχείο ύψης της σημασίας για το μέλλον μας. Όμως παράλληλα τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η ΕΠΑ και η ΚΕΠΑ δεν είναι εθνικές πολιτικές, είναι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ε, θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ελέγχουν αυτές τις διαρθρώσεις. Έχουμε εκλεγεί άμεσα από τους Ευρωπαίους πολίτες και γι' αυτό ακριβώς η συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων αλλά και του Ευρωπαϊκού. Γι' αυτό ακριβώς ο κοινοβουλευτικός έλεγχος θα πρέπει να ασκηθεί και από το δικό μας σώμα και από τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει μια ε, νέα καινοτόμο δομή για την νομιμοποίηση της ε, ε, δημοκρατικής, της ευρωπαϊκής, των ευρωπαϊκών δημοκρατικών δρόμενων. Γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί μία νέα ισότιμη διάρθρωση. Αυτό δεν το προβλέπει όμως η συνθήκη της Λισαβόνας και όπως υπενθύμησαν πολλοί, θα ήταν σκόπιμο να τονίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό ε, διαδραματίζει κέριο ρόλο. Η δυνάμη του άρθρου 37. Έλεγχο της ΕΠΑ και της ΚΕΠΑ και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, διαδραματίζει ένα νέο ρόλο όπως ε, τόνισε και ο Άντριου Νταφ. Γιατί μιλάμε για στρατιωτικές και πολιτικές ικανότητες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η καινοτομία. Είτε δεν θα συνεννοηθούμε και ο καθένας θα ακολουθήσει το δρόμο του, και δεν θα ερμηνεύσουμε σωστά το πρωτόκολλο ή θα βρούμε τη σωστή διάρθρωση διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. με βάση θεσμούς και θεσμικά όργανα που το καθένα διατηρεί τις δικές του δομές. Άρα δεν μιλάμε για νέα γραμματεία. Μιλάμε για νέες δομές εποπτείας. για να προασπίσουμε έναν πραγματικό διάλογο. Θα πρέπει λοιπόν να εξεύρουμε τα κατάλληλα μέσα συνεργασίας, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε, να ακολουθήσουμε διαφορετικό δρόμο. Κύριος Σουκάρσκι από την ε, Βουλγαρική Βουλή. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να λάβω μέρος σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτό το διάλογο. Γνωρίζω ότι έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας, κανονικά θα πρέπει τώρα να έχουμε πάει για το γεύμα, αλλά οπωσδήποτε η ικανότητα παρακολούθησης ε, των παρισταμένων έχει ασφαλώς μειωθεί και γι' αυτό θα προσπαθήσω να περιοριστώ στα τρία λεπτά. Η πολιτική άμυνας είναι η λιγότερο κοινή πολιτική σε σχέση με την ΚΕΠΑ και θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι εννοώ. Οι χώρες, τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν το ποσοστό κυριαρχίας που μπορούν να διεκδικήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει από μόνη της στατιωτικές δυνάμεις. και γι' αυτό το λόγο απαιτείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος από τα εθνικά κοινοβούλια. Όταν μιλάμε για κοινοβουλευτικό έλεγχο, θα ήθελα να πω πώς διεξάγεται αυτός ο έλεγχος από τα εθνικά κοινοβούλια. Ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν είναι εναρμονισμένος σε οικουμενικό επίπεδο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κοινοβουλευτικό έλεγχο που να λαμβάνει υπόψη την πολυμέρεια που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλίων. Πρέπει να, ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που υπάρχουν από κοινοβούλιο σε κοινοβούλιο. Είναι ευτυχές γεγονός ότι η σύσταση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί κάποιο χρόνο που θα μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε ορισμένα στοιχεία της ΕΠΑ. Οι διπλωμάτες όταν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους θα έχουν, ελπίζω, μία ουσιαστική σαφώς καθορισμένη πολιτική πάνω στην οποία θα στηριχθούν, η οποία πρέπει να υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και Ζητώ από τους εθνικούς βουλευτές να επιταχύνουν τη διαδικασία διαλόγου στο πλαίσιο των εθνικών κοινοβουλίων ώστε να εφαρμοστεί σε κοινοτικό επίπεδο ένα ικανοποιητικό σύστημα κοινοβουλευτικού ελέγχου που θα επιτρέψει να, στους ε, εθνικούς βουλευτές να αναλάβουν τις αρμοδιότητες τους. Ο κύριος Ομήρου παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Ανταποκρίνομαι στην έκκλησή σας να είμαι σύντομος. Έχω ορισμένε σύντομες παρατηρήσεις συνοπτικά. Η συνθήκη της Λισαβόνας πράγματι προσφέρει νέες ευκαιρίες σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη τόσο της ε, ΚΕΠΑ, κοινή εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, όσο και της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Θέλω να σημειώσω το εξή ότι για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ορατό ρόλο στην διεθνή πολιτική σκηνή, χρειάζεται να προωθήσουμε και να εμβαθύνουμε αυτές τις πολιτικές. Παρατήρηση δεύτερη. Εκ των όνου κάνευ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που σύμφωνα με τη συνθήκη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ΚΕΠΑ. Παρατήρηση τρίτη. Δεν μπορεί βεβαίως να υπάρξει κοινοβουλευτικός έλεγχος χωρίς τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, αφού πρόκειται για πολιτικές που εμπίπτουν στην διακρατική σφαίρα. Η εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι απαραίτητη, αφού είναι τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, αρμόδια και υπεύθυνα για τον έλεγχο των εθνικών πολιτικών άμυνας είτε σε ό,τι αφορά τις σχετικές αποφάσεις πολιτικής, είτε σε ό,τι αφορά την αποδέσμευση των σχετικών κονδυλίων. Παρατήρηση τέταρτη, η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι και θεμητή και απαραίτητη, κυρίως λόγω της εξειδίκευσής του στην ευρωπαϊκή διάσταση των πολιτικών ε, αυτών, αλλά και της συνεργασίας και της τριβής του Κοινοβουλίου με τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς, όπως είναι η ύπατος εκπρόσωπος για θέματα εξωτερική πολιτικής και πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Άρα λοιπόν, μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας συνδυάζει διακρατικό και κοινοτικό έργο, διτής φύσης συνεπώς πρέπει να είναι και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Και μια παρέκβαση με την άδεια σας. Θέλω να χαιρετήσω τις παρεμβάσεις συναδέλφων στην συζήτηση του προηγούμενου θέματος για την ανάγκη λύσης του Κυπριακού για να πάψει αυτή η ε, δημιουργία προβλημάτων και δυσχεριών σε ό,τι αφορά την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ο Κύπριος συνάδελφος μου, ο κύριος Νεοφίτου, έδωσε ήδη ικανοποιητικά, κατά τρόπο πολύ ορθό, τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ήθελα απλώς να σημειώσω το εξής. Δεν είναι αρκετό να υπάρχουν θεωρητικού χαρακτήρα προσεγγίσεις και ε, ευχολόγια για τη λύση του Κυπριακού και θέλω να επισημάνω και τις ευθύνες και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποσύρουν αυτό τον λεγόμενο κανονισμό για το απευθείας εμπόριο που αν πραγματικά υιοθετηθεί σας λέω με κάθε ειλικρίνεια τελειώνω θα υπάρξει θανατηφόρο πλήγμα σε, στις προσπάθειες λύσης του κυπριακού προβλήματος. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ήδη έχουμε καθυστερήσει δεν είναι μόνο για το δικό μας γεύμα, έχουμε και κάτι διερμηνείς που εργάζονται και είναι πάρα πολλοί και ε, δέχτηκαν να παρατείνουν κατά λίγο να κάνουν υπέρβαση του ωραρίου. Παρακαλώ σεβαστείτε και το δικό τους ωράριο και τη δουλειά τους. Ο κύριος Ζιγκέρης, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Λιθουανικής Βουλής. Ε, Στα γερμανικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον φίλο μας ε, κύριο Μπροκ και αγαπητοί συνάδελφοι Ε, ε, τον ευχαριστώ ε, πραγματικά και για το ρόλο του. Ε, θα πρέπει να πούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι πρεσβεύουμε. Έχουμε ένα σύστημα αξιών και αρχών που ευαγγελιζόμεθα. Δεν είναι μια απλή ήπειρος, μια κάποια ήπειρος η Ευρώπη. Έχει και μια ιστορία η Ευρώπη. Με δύο παγκοσμίους πολέμους στον 20ο αιώνα. Έχουμε μια ιστορία ε, ε, με τη Γαλλική Επανάσταση, τη Γαλλική ε, Ρεπιμπλίκ και αυτό σημαίνει ότι κυριαρχεί το κοινοβούλιο. Η κοινοβουλευτική διάσταση έχει την κυριαρχία και αυτό είναι εγγύηση αξιών και αρχών. Εμείς έχουμε τρεις επιτροπές από τη Βουλή μας και τρεις προτάσεις ε, η πιο απλή είναι η εξή. Ε, είπατε ότι ε, θα θέλετε να συστηθεί μια συνέλευση κόφακ. Αλλά εκεί θα πρέπει να συμμετέχουν και οι ε, συνάδελφοι της άμυνας. Να μην έχουμε κόφακ και κόντακ που είναι και δυσάρεστα τα αρχικά τους, να είναι κόφντακ που ακούγεται καλύτερο και δεν έχει και επιπλέον κόστος. γιατί δεν έχουμε δύο δομές. Αυτή είναι η πρότασή μας της λιθωνικής πλευράς. Ε, και εκεί θα είναι οι ε, εκπρόσωποι από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από άλλους συναδελφούς γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τον Άτο. Είναι σύμμαχος, είναι ε, εταίρος και έτσι θα έχουμε και καλύτερη αξιοποίηση ε, των οικονομικών πόρων. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε, επαναλαμβάνω, καλύτερη διαχείριση των οικονομικών, πιο ορθολογική χρήση, ενημέρωση, συνεννόηση και θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Μπορεί να είμαστε ε, και λιγότερο δημοφιλείς στη χώρα μας βέβαια όταν μιλάμε για αμυντικούς προϋπολογισμούς. Ο κύριος Γκάλερ από πλευράς του ΕΛΚ που δεν μίλησε ακόμα το ΕΛΚ πάρα πολύ γρήγορα και ο Μπρόκ για να κλείσει. Ευχαριστώ. Άκουσα πολλούς συναδέλφους στο Εθνικό Κοινοβουλίο και νομίζω ότι φοβούνται μήπως χαθεί η κοινή τους εμπειρία που έχουν αποκομίσει από τη, ΒΕ, από τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή δεν έχουμε εμεί τέτοια πρόθεση, ούτε τέτοιο συμφέρον. Το είπε και ο κύριο Μπρόκ στην αρχή. Θα συναντιόμαστε τακτικά και θα συζητούμε για συγκεκριμένα θέματα, όχι πανηγυρικέ συνεδριάσει γενικά και αόριστα ομιλίε, για συγκεκριμένα θέματα. Παράδειγμα, να συζητήσουμε μία ε, αποστολή εξωτερική. Εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να συμφωνήσουμε για το πολιτικό σκέλος, γιατί είναι στη δική μας αρμοδιότητα. Και εσείς, στα Εθνικά Κοινοβούλια, μπορείτε να συμφωνήσετε με το στρατιωτικό σκέλος του αμυντικού προϋπολογισμού, γιατί είναι δική σας αρμοδιότητα σε αυτή λοιπόν τη συγκεκριμένη περίπτωση ας εξετάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε απέναντι στην εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Αυτό όμως που δεν γίνεται κατά την άποψή μου είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο νομιμότητες που υπάρχουν που είναι ευρωπαϊκή νομιμότητα και εθνική νομιμότητα δεν μπορούμε να βάλουμε σφήνα τώρα ένα τρίτο επίπεδο γιατί ε, μετά δεν μπορούμε να συνδυάσουμε, να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας. Η Βουλή των Κοινοτήτων ποτέ δεν πέρασε ε, ομόφωνο ο ψήφισμα της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης ε, από τη Βουλή. Δεν το, δεν το θεώρησε δηλαδή δεσμευτικό ακόμα και αν ήταν ομόφωνο. Και αν είχαν ψηφίσει στη ΔΕΕ οι Βρετανοί συνάδελφοι. Η ε, νομιμότητα είναι εθνική υπόθεση και δεν είναι σε μια ακόμα συνέλευση. ε, γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που προτείνει ο κύριος Μπροκ να έχουμε τακτικές επαφές και συνεδριάσεις ε, για συγκεκριμένα θέματα. Ε, είναι σωστό. Και για τη γραμματεία που ζητάτε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε όλες τις δυνατότητες. Και εσείς ε, ως εθνικοί βουλευτές έχετε όλοι γραφεία στις Βρυξέλλες και οι συνάδελφοι, οι υπάλληλοι που είναι στα γραφεία του Κοινοβουλίου και στις δικές τους αντιπροσωπείες μπορούν να συνεργάζονται με τις δικές μας δομές για να προετοιμάζουμε τα πάντα όπως πρέπει και προς αμοιβαίο συμφέρον. Ευχαριστώ. Ο Έλμαρ για να μας ε, πει ορισμένα συμπεράσματα από αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας, διότι διευκρινίστηκαν στο μυαλό μου κάποια θέματα και από αυτά που άκουσα. Να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφος Γκάλερ. Ο καθένας θα πρέπει να εκτελεί το έργο του με βάση αυτά που ορίζει το σύνταγμά του. Και δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε σε ένα οποιοδήποτε θεσμό που δεν προβλέπεται πουθενά. Αν θέλανε ξεχωριστό κοινοβούλιο για την ΚΕΠΑ θα το είχαν γράψει στη συνθήκη. Δεν το κάνανε όμως και γράψανε συνεργασία. Αυτό δεν σημαίνει έλεγχος αλλά ανταλλαγή απόψεων. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να υπάρχει και συνέχιση ε, της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει να πάρουμε τη σκητάλη. Ποια σκητάλη, εγώ δεν βλέπω καμιά σκητάλη που θα πρέπει να συνεχίσουμε εμείς, τη ΔΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, ε, υπερασπίζεται τα δικαιώματά του όπως θα τα υπερασπιστεί και το κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο βάσει των συνθήκων και βάσει των συνταγμάτων. Και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Κάτι άλλο που ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε και το προσφέρω Κάποιο είπε ότι υπάρχει ένα μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα μετά τη Λισαβόνα. Ούτε αυτό το έλλειμμα το βλέπω. Και αν υπάρχει, να το εξετάσουμε. Και σα προτείνω από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σα στείλουμε ένα έγγραφο και να κάνουμε έρευνα. Πού βρίσκονται οι αρμοδιότητες και πού ενδεχομένως να υπάρξει έλλειμμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Γιατί μπορεί και να σφάλω, δεν ε, λέω. Να το συζητήσουμε και αυτό αν διαπιστώνουμε, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε τέτοιο έλλειμμα, να κοιτάξουμε πώς θα το κλείσουμε. Μέχρι τώρα δεν είπε κανείς συγκεκριμένα πού είναι το έλλειμμα. Καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε και συνείδηση των δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά ε, τη συνδίκη της Λισαβόνα και μετά τις διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα πρέπει να τα ξαναπούμε σε λεπτομέρειες για να δούμε και τις συνέπειες. Πρόταση ακούω τώρα για Κόζακ θα είναι επιτροπές ευρωπαϊκών υποθέσεων. Όχι ούτε εξωτερικών, ούτε αμήνης. Κατά τα άλλα, σας είπα ποια δικαιώματα έχουμε σε κάποιους τομείς. Και το θέμα δεν είναι από τη μια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την άλλη όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν καταλαβαίνω γιατί και από πού το βρίσκεται από τη συνθήκη της Λισαβόνα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι το 1,28 δηλαδή 27 κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με ίση εκπροσώπηση. Και το Κοινοβούλιο όταν βλέπει ε, ε ότι υπάρχουν επεμβάσεις στα χωράφια του, στις αρμοδιότητες, τι θα κάνει.